Um, λοιπόν, συνάδελφοι, έχει πάει σχεδόν 9 ε, ναι και 10 και όπως ξέρετε έχουμε και τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια οι οποίοι θα έρθουν στις 9.30 για μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση για να συζητήσουν τους ε, στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και την ε, ανάπτυξη ε, και έχουμε και μέλη από τις Επιτροπές Ελέγχου για την Ανάπτυξη από 24 κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνεδρίαση. Όπως βλέπετε έχουν προσκληθεί πολλοί συνάδελφοι. Έχουμε και καλεσμένους από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, από αρκετές αφρικανικές ε, χώρες. Ελπίζω λοιπόν να παραμείνετε λοιπόν και να τους ακούσετε, διότι θέλουμε να δούμε πώς εφαρμόζουν οι ίδιοι τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, θα δούμε και τι κάνουν τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Κάθε χρόνο ε, οι χώρες υποβάλλουν έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη και ε, αναφέρουν τις επιδόσεις τους. Και φέτος ε, το Ίδρυμα θα μας παρουσιάσει μια εικόνα του τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα πάει στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν πρόγραμμα με τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, από τις 9.30 μέχρι τις 12.30 και ελπίζω οι συνάδελφοι να μείνουν για να ε, παρακολουθήσουν αυτή την τόσο σημαντική συνεδρίαση. Στην ε, αρχή της χθεσινής συνεδρίασης είπα ότι είναι Αφρικανική εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Πολλά συμβαίνουν. Απόψε υπάρχει μία ομάδα για την υποστήριξη της δημοκρατίας και τις εκλογές στην Αφρική, στις 14 ε, και 45 και ο πρόεδρος αύριο διοργανώνει μια μεγάλη διάσκεψη ε, για την Αφρική με πολλές αφρικανικές χώρες. Υπάρχουν αφήσει σε όλο το κοινοβούλιο, έχετε προσκληθεί σε αυτή τη διάσκεψη, έχετε προσκληθεί να δείτε, ε, να μιλήσετε σε αυτή τη διάσκεψη και ελπίζω να συμμετέχετε όλοι. Έχουμε δύο ψηφοφορίε όμω πριν περάσουμε στην συνεδρία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Καταρχά να κάνουμε έναν έλεγχο για να δούμε ότι λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Σα παρακαλώ πατήστε το κουμπί σα. Ο κύριο ε, Λέντα πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μπορείτε να περιμένετε δύο λεπτάκια, διότι μόλι με ενημέρωσαν συνάδελφοι που έρχονται, υπάρχει, είναι εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι μέλη τη Επιτροπή. Με συγγνώμη για την... Ο κύριο Ρούμπι και ο κύριο Τσέλερ. Ναι, να περιμένω. αλλά έχει πάει και 9 και 10. Ένα λεπτό ακόμα θα περιμένουμε. Διότι δεν είναι σωστό για του υπολείπου. Υπάρχουν και πολλοί από την άλλη πλευρά που δεν είναι εδώ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε 10-15 λεπτά γιατί δεν έρχουν. Ελπίζω να επιδείξετε λίγο πνεύμα συμβιβασμού, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, τουλάχιστον να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ, πατήστε το κουμπί σας. Υπάρχει ούτως ή άλλως τεχνικό πρόβλημα, επομένως πρέπει να επιλύσουμε πρώτα το τεχνικό πρόβλημα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Πρέπει να διακάψουμε μισό λεπτό. We have the um, here on the screen. Έχουμε εδώ αποτέλεσμα ψηφοφοριών στην οθόνη, αλλά δεν βγαίνουν στην κεντρική οθόνη ε, μιλήσετε με τον τεχνικό να επιλύσουμε τα τεχνικά προβλήματα. On your screen as well in front of you. Τα έχετε και εσείς στην οθόνη σας ούτως ή άλλως, οπότε μπορείτε όλοι να δείτε το αποτέλεσμα. Δεν μπορείτε. Για να ξαναδοκιμάσουμε. Πατήστε όλοι το κουμπί σας. Δεν υπάρχει σήμα στις οθόνες. Για να μην no signal. Πέρασε της ψηφοφορίας. Ναι, εγώ έχω τα αποτελέσματα, εσείς τα βλέπετε στις οθόνες σας. Ωραία. Επομένως μπορείτε να δείτε και εσείς τα αποτελέσματα και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ζητώ συγγνώμη Μπόγκταν, αλλά είναι σχεδόν 9 ε, και 4 και 9.30 έχουμε τις συνεδρίες. Θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Πρώτα λοιπόν, είμαστε στο σημείο 9, ισότητα των φίλων στις εμπορικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης ήταν η Λόλα Σάνσες. Λόλα, θέλεις να πεις κάτι πριν ψηφίσουμε? Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε απευθείας. Και ξεκινάμε. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της Εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 35, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 ψήφι κατά, 10 υπέρ, μία αποχή. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της συμβαστικής τροπολογίας 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά είναι δύσκολο να παρακολουθώ γιατί δεν υπάρχει κανεί στη μέση. Τροπολογία 48. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάντα την ίδια πλειοψηφία έχουμε. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 57, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση της 58 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση της 59 άρχεται η ψηφοφορία Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα δούμε. Πέρα τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αλλά ήταν πολύ κοντά. 60 υπέρ, κατά, επαλήθευση της 60, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, επαλήθευση 63, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 64 υπέρ, υπέρ, επαλήθευση 64, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ελέγχουμε την 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση της 4 νομίζω ότι εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε της ψηφοφορίας. Καταπίπτει. Απορρίπτεται μάλλον για την 11-11 το αποτέλεσμα. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της προφορικής τροπολογίας 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και πάλι. Ισοψηφία. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση της 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ. Επαλήθευση της 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Επαλήθευση της 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Ελέγχουμε και τη 15. Ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Επαλήθευση και τις 16, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με μία ψηφοδιαφορά Ψηφίζουμε το σχέδιο γνωμοδότησης ηλεκτρονικά με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κάποιος έχει την κάρτα του, αλλά δεν ψηφίζει. Αν το κάνετε από επιλογή, εντάξει. Αν θέλετε όμως να σας καταγράψουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ πατήστε το κουμπί. Αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα εάν κάποιο δεν έχει ψηφίσει σωστά. Πέραση τη ψηφοφορίας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στη Λόλα Σάνσες. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 10, μια ακόμα γνωμοδότηση. για την Επιτροπή Γυναικών. επί της ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή Γυναικών. Συντάκτης γνωμοδότησης, ο κύριος Μαρτσελέση, θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω απλά να πω ότι την ε, προηγούμενη εβδομάδα ενεκρίθη το πρώτο σχέδιο δράσης ε, με σχέση, σε σχέση με το φίλ για την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για το θέμα αυτό. Μετά τη Βόνη νομίζω πλέον έχει καταστήσει σαφές ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε εδώ τη δουλειά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω όλοι να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Αυτά είχα να πω για την COP23 στη Βόνη. Ωραία, τροπολογία είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική α, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6, ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέξουμε τροπολογία 6, άρχεται ψηφοφορία. Νόμιζα ότι έχει καταπέσει Μαρία, έχει καταπέσει, καλύπτεται από τη συμβαστική. Πάμε στην 6 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6. Ξεκολουθεί να είναι ανοιχτή η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Μισό λεπτό. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία. δεν ε, τα κάναμε σωστά. Ξανά αρχίζει η ψηφοφορία τροπολογία 6. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορία. Δεν το βλέπω. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Λοιπόν, πηγαίνουμε στην τροπολογία 7, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 7, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται σαφώς. Πέρασε ψηφοφορία, δεν το κατάλαβα, λοιπόν, πρόεδρο, συγγνώμη. Τώρα το βλέπω. Έχει απορριφθεί, σαφώς. Συμβιβαστική K, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, ψήφι υπέρ. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Καταπίπτει. Πηγαίνουμε στη συμβαστική B. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 15. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική C. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε τη 18 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 20 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ όχι λάθος. Συγγνώμη. Έχει καταπέσει. Συμβαστική E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31, ψήφι υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε την 31, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Συμβιβαστική G, ψήφι υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Έλεγχος για 35. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H ψήφι Κατά ποχέ εγκρίνεται. Τώρα, η τροπολογία 38, ψήφι υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε την 38, άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τώρα πρέπει να πάμε στην 43. Όχι, μισό λεπτό. 38 δεν έγινε δεκτή. 39 wasn't adopted, right. Θα πάμε στη 39 από ό,τι φαίνεται. 39 ψήφι υπέρ. Τη 39. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα, που πάμε, στην 43. Ψήφι υπέρ. Κατά, Απορρίφθηκε. 44 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε τις 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Μπορεί και να εγκρίθηκε αλλά δεν είμαι σίγουρη. Πέραση ψηφοφορίας. Πράγματι εγκρίθηκε. 46 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική I ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται. Και αλλάζουμε σελίδα, πηγαίνουμε στην συμβαστική J. Ψήφι περ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55, ψήφι Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57, ψήφι περ Κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε την 57, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τώρα πηγαίνουμε στην 58. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Τι θέλετε. Ο Ερνικέ Γκερέρο κάτι θέλει να πει για την τρόπο 60. Θέλω να την αποσύρω την 60 λέει ο κύριο Γκερέρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αποσύρεται 60, πηγαίνουμε στην 61. Ψήφι υπέρ. Κατά απόχε, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε συνολικά την γνωμοδότηση ω τροποποιήθη και ονομαστικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Μαρσελέση. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Κάνουμε εδώ μία διακοπή της συνεδρίασης γιατί στη συνέχεια έχουμε την συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και θα αλλάξει το setting εδώ. Okay, colleagues, we're going to make a start. So if everybody could take their seats. Λοιπόν, συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε την πρωινή μας συνεδρία με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έπρεπε να περιμένουμε τους καλεσμένους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια και από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο έπρεπε να βρουν το, την αίθουσα και αυτό δεν είναι πάντα εύκολο σε αυτό το λαβύρινθο εδώ. Λοιπόν, εκ μέρου τη Επιτροπή Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω τη χαρά να καλωσορίσω όλου του συναδέλφου στη σημερινή μα ε, συνάντηση. Θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων μαζί σα, την οποία θεωρούμε πολύ ε, σημαντική εμεί και ελπίζουμε και εσεί να την βρείτε ενδιαφέρουσα. Θα συζητήσουμε για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση από την δική μα πλευρά του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εφαρμόσει αυτού του στόχου μέσω τη ε, πολιτικής, της εξωτερική πολιτική τη. Έχουμε, γνωρίζω ότι πολλοί από εσά ε, προέρχεστε από τι επιτροπέ εξωτερικών των κοινοβουλίων σα. Αλλά είναι γιατί είναι και αυτός ε, ένας, μια πτυχή, είναι γι' αυτό μια πτυχή της εφαρμογής των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης πέρα από την εθνική εφαρμογή τους. Γιατί ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε οι δικές μας πολιτικές, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εθνικές πολιτικές, να εξυπηρετούν, να εξυπηρετούν αυτούς τους στόχους. Σήμερα όμως θα σταθούμε στην εξωτερική διάσταση. Ονομάζομαι Λίντα Μακαίβαν, είμαι ε, πρόεδρος της Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν μέλη από πολλές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από, πολιτικές, ε, από πολλές πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερως ευτυχής για την παρουσία σας εδώ και ελπίζω να βρείτε την συζήτηση τη σημερινή χρήσιμη για εσείς. Να σας ενημερώσω ότι πέραν από τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων έχουμε και εκπροσώπους από, από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η, οποία είναι εκείνη που ε, επιβλέπει την εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Έχουμε επίσης εκπροσώπους από το Πέλτερμαν Stiftung και από το Sustainable Development Solutions Network, δύο οργανώσεις οι οποίες θα μας ε, κάνουν κάποιες παρουσιάσεις εκπρόσωποι τους στο δεύτερη ε, συζήτηση, στο δεύτερο πάνελ. Θα συντονίσω εγώ το πρώτο μέρος της συζήτησης και η κυρία Θεοχάρου στο δεύτερο. Κάποιες πρακτικές ε, παρατηρήσεις, θέματα για τα οποία πρέπει να σα ενημερώσω. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο ίντερνετ, μέσω streaming, επομένως εάν κάποιος στο, στη χώρα καταγωγής σας το επιθυμεί θα μπορούσε να τη δει ζωντανά στο ίντερνετ ή και αργότερα. Υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό των Ολλανδικών, των Σλοβενικών, των Μαλτέζικων, των Λετωνικών και των Γεδελικών. Μπορείτε να βρείτε στον ε, πίνακα στην οθόνη ε, το κανάλι στο οποίο μπορούσε να, μπορείτε να ακούσετε την διερμηνία την δική σας γλώσσα. Τα ελληνικά βρίσκονται στο κανάλι 7. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να ζητούν το λόγο απλώς σηκώνοντας το χέρι τους, ε, ως συνήθως. Τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων που επιθυμούν να λάβουν το λόγο, ε, θα ήθελα να σας ζητήσω να συμπληρώσετε ένα καρτελάκι, μια μικρή φόρμα που υπάρχει στο έδρανό σας, και να το δώσετε σε κάποιον από τους ε, κλητήρες της αίθουσας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε το όνομά σας και να σας δώσω το λόγο. <clears throat> Ναι, οι κλητήρες θα το φέρουν στο Προεδρείο. Επομένω, το συμπληρώνετε, το σηκώνετε και ένας κλητήρας θα το φέρει στο, στο Προεδρείο. Και αυτό σας το ζητώ επίση για να φροντίσουμε να δοθεί επαρκής χρόνος ομιλίας σε όλους... Αν το γνωρίζετε ήδη ότι επιθυμείτε να λάβετε το λόγο, σας παρακαλώ συμπληρώστε από τώρα αυτή τη φόρμα για να ε, σχεδιάσουμε καλύτερα τη συζήτηση. Θα ξεκινήσουμε με παρουσιάσεις και με μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εφαρμόσει την κοινή αντίληψη για την ε, ανάπτυξη. Και το δεύτερο σκέλος της συνεδρίασής μας θα ε, το αφιερώσουμε στον τρόπο με τον οποίο εσείς, οι διάφορες χώρες, σκοπεύουν να εφαρμόσουν τους στόχους αυτούς μιας και έχουμε πολλούς ομιλητές, θα πρέπει να περιορίσουμε το χρόνο ομιλίας αυστηρά σε δύο, δυόμιση, ακόμα και ένα λεπτό και θα σας ενημερώνω όταν θα εκπνέει ο χρόνος ομιλίας. Σας παρακαλώ να τον κηρύτε για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. <clears throat> θα ήθελα να ξεκινήσουμε με με ένα, βλέποντας ένα ε, βίντεο Ε, η οποία είχε, το οποίο ε, το τραβήξαμε σε μια εκδήλωση την οποία είχαμε οργανώσει από κοινού με τα Ηνωμένα Έθνη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Ηνωμένα Έθνη, για την ε, ημέρα βιώσιμη ανάπτυξη. The Sustainable Development Goals are an ambitious agenda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 Well, Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό το βίντεο το παρήγαγαν τα Ηνωμένα Έθνη στην εκπρόσωπο με τον οποίο σύντομα θα δώσω το λόγο. Θα ήθελα να, βοηθήσω, να, να ε, ευχαριστήσω μάλλον την κυρία Ρίτς, μια συνάδελφο η οποία βοήθησε ε, πολύ στην διοργάνωση της, της σημερινής εκδήλωσης. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει ένας φωτογράφος και μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους ε, στόχους τους, ε, της βιώσιμης ανάπτυξης και να φωτογραφηθείτε μπροστά από ένα σχετικό ε, πλακάτ για να δώσετε μια κάποια δημοσιότητα, επιλέξτε ποιο θα θέλετε, ποιον στόχο, ποιον στόχο θα θέλετε να σταθείτε. Στις 12 και 20 θα γίνει αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μπάρμπαρα Πέσε Μοντέιρο, διευθύντρια του Γραφείου Ρεξελών, του Προγράμματος για την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, η οποία θα ξεκινήσει τη συζήτησή μας. Ε, έχει υποστηρίξει με όλες τις δυνάμεις την ε, υιοθέτηση και την προσπάθεια να επιτύχουμε τους βιώσιμους στόχους της χιλιετίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήξερα ότι θα δείξετε αυτό το βίντεο. Εκεί λέγονται πολλά σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω και εγώ και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και νομίζω ότι μεγάλο μέρος ε, της δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην παραμείνει αυτή μια συζήτηση μεταξύ πυρογνωμόνων, αλλά να καταστεί πολιτική συζήτηση και να κινητοποιηθούν οι διάφοροι φορείς και παράγοντες που πρέπει να συμμετέχουν στην προσπάθεια και μάλιστα πρέπει να προχωρήσουμε με ταχύς ρυθμούς. Φαντάζομαι ότι θα έχετε τη δυνατότητα να το συζητήσετε, όμως το θεματολόγιο αυτό αφορά και τον ιδιωτικό τομέα και τις ε, τοπικές αρχές και για τα εθνικά κοινοβούλια όπω θα αναφέρω. Το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια κάθονται στο δύο τραπέζι για να συζητήσουν το θεματολόγιο αυτό, πραγματικά δίνει μεγάλη δύναμη στην όλη προσπάθεια. Και είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα, διότι ολοκληρώθηκε η COP23 για το κλίμα και αυτό νομίζω υπογραμμίζει το γεγονός ε, του πόσο επίγον είναι αυτό το θεματολόγιο. Και δεν μπορούμε να το αναβάλουμε συνεχώς ή να το αφήνουμε για τις επόμενες γενιές. Είναι κάτι που μας αφορά καθημερινά και δεν αφήνει κανέναν εκτός. Συνοπτικά. Για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης φαντάζομαι ότι γνωρίζετε, αλλά το θέμα είναι να μην μείνει κανείς πίσω και πουθενά. Άρα πρόκειται για ένα θεματολόγιο. Εγώ βέβαια θα μιλήσω πιο πολύ για την εξωτερική συνιστόσα του θεματολογίου. Εσείς είστε εθνικοί βουλευτές και ευρωβουλευτές και εδώ το θέμα είναι ο απλός κόσμος. Το είπα και στην ε, παρουσίαση στο βίντεο. Δεν θέλουμε να μείνει κανείς εκτός των εθνικών πολιτικών και όλοι θέλουμε να ωφεληθούν από την ανάπτυξη. στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι κάποιες λέξεις που δεν λένε και πολλά, αλλά είναι παγκόσμιοι ε, οι στόχοι και αφορούν όλες τις χώρες ε, του πλανήτη, όχι μόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο της συζήτησης που θα γίνει στην Ευρώπη, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ θετικό θεματολόγιο να συζητήσουμε. Μιλάμε για βιώσιμη κατανάλωση, βιώσιμη παραγωγή, αλλά και για βασικά δικαιώματα. Μιλάμε για τους νέους, τις νεαρές γυναίκες, τον άνθρωπο και αφορά πολλά ζητήματα που μας ενδιαφέρουν στις χώρες μας. Για παράδειγμα, απασχόληση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερη μετανάστευση προς την Ευρώπη, όπως είπε και ένας βουλευτής, αλλά είναι και ένα ισχυρό θεματολόγιο γενικά για την Ευρώπη. Αν λοιπόν καταφέρουμε να δεσμευτούμε και με αφοσίωση και οικοδομητικά για το θεματολόγιο και να μην συζητάμε μόνο για τα προβλήματα, αλλά προωθούμε ένα θετικό όραμα για το μέλλον και με συγκεκριμένο διάγραμμα θα πετύχουμε πολλά. Είναι ένα θεματολόγιο βέβαια πολύ φιλόδοξο. Ίσως υπερβολικά φιλόδοξο είπαν ορισμένοι. Νομίζω ότι είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Είδαμε και στη Βόνη και στις συζητήσεις για τη Συμφωνία των Παρισίων ότι υπάρχει ανάγκη για φιλοδοξία στον τομέα αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε τι θα πει και πρέπει να εμψυχώσουμε, να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες όπου και δραστηριοποιούνται. Εγώ βρίσκομαι εδώ και εργάζομαι στις Βρυξέλλες και έρχομαι και συχνά στο Κοινοβούλιο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώ δηλαδή για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά μιλώ και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε εσείς να είστε ηγέτες, ε, οι πρωτοπόροι, μέσω των συμφωνιών που επιτυγχάνετε και μέσω της εφαρμογής των συμφωνιών αυτών. Πολλές από τις μεγάλες συμφωνίες πολλές φορές δεν θα μπορούσαν να βγουν από το πλαίσιο των ΗΕ ή ούτε καν να ε, εγκριθούν αν δεν υπήρχε υποστήριξη των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Άρα μιλάμε για στρατηγική εφαρμογή, στρατηγική υλοποίηση. Η συνένεση επίσης είναι κάτι θετικό, το consensus, τα πει ο Κάσπαρ στη συνέχεια. Πρόκειται για μια δέσμευση της Ένωσης ε, για την υποστήριξη της αφαρμογής των στόχων για τα επόμενα 15 χρόνια στις χώρες εταίρους. Έχουμε συνεισφέρει τα μάλλα σε αυτή την προσπάθεια. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ισχυρή. Και αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλα τα στοιχεία, τα προγραμματικά του προγράμματος. Τόσο να δούμε πώς μπορούμε στρατηγικά να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση. Γιατί επί τόπου όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Μπορεί να το γνωρίζετε, έχουμε μεταρρύθμιση αυτή την εποχή ε, στα Ηνωμένα Έθνη, γιατί θέλουμε να προσαρμοστούμε ε, στις εξελίξεις για να μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε το θεματολόγιο 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, που δεν αφορούν πλέον τομείς, υπάρχει αλληλεπίδραση όλων των σχετικών αυτών τομέων. Αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους, χάρη να μειώσουμε τη φτώχεια, που είναι ο πρώτος στόχος, θα πρέπει να δούμε τις ανισότητες ή και τα θέματα του φύλου. Το είπε και κάποιος στο βίντεο, αν θυμάστε. Επίσης, οικονομική ανάπτυξη. Δεν μπορεί κανείς απομονωμένα από τους θεσμούς να αντιμετωπίσει τα σχετικά ζητήματα. Αυτή είναι η προσέγγιση λοιπόν Μπορεί και να μην είναι βέβαια το θέμα του πρώτου πάνελ, της πρώτης συνεδρίας, ωστόσο θα επιμείνω και θα τονίσω ότι θα πετύχουμε μόνο αν συμμετέχουν όλοι και αν δείξει η ηγεσία η Ευρώπη όσον αφορά την εξωτερική συνιστόση. Αν εφαρμοστούν οι στόχοι δηλαδή στην Ευρώπη πρώτα απ' όλα. Και θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την ε, πλατφόρμα των πολλών ε, εμπλεκομένων multi-stakeholder platform. Υπάρχει εξωτερική, εσωτερική συνιστόσα και τα μηνύματα που έχουν δοθεί είναι πολύ θετικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και τα κράτη-μέλη δεν κάνουν από τη δική τους πλευρά προσπάθειες που έρχονται να συμπληρώσουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τον Ιούλιο είδαμε τις εκθέσεις, ε, τις εθελοντικές εκθέσεις πολλών ευρωπαϊκών κρατών, κρατών είναι οι περισσότερες που έχουν ε, υποβάλει τέτοιες εκθέσεις. Το Βέλγιο, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αύριο θα έχει μια πάρα πολύ ευρεία ε, συνάθρηση που θα παρουσιάσει την έκθεση στην βελική κοινωνία, στην νεολαία, στη κοινωνία των πολιτών, στις τοπικές αρχές και θα παρουσιάσει και ένα σαφές πρόγραμμα υλοποίησης για τις δημόσιες πολιτικές, για παράδειγμα, για το προϋπολογισμό, και τομέα κτλ. Για να κινητοποιηθούν όλοι αυτοί και να εφαρμόσουν τις ίδιες ε, διαδικασίες, ατενίζοντας το μέλλον. Πολλά έχουν γίνει μετά την ε, Συμφωνία επί του Θεματολογίου. Κάθε Ιούλιο, είπαμε, έχουμε αυτές τις εκδηλώσεις και εθελοντικά οι χώρες παρουσιάζουν ε, τις ε, επισκοπήσεις τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δείχνει πως οι χώρες έχουν την κυριότητα αυτής της διαδικασίας, την έχουν ιδιοποιηθεί και δεν μιλάμε πλέον στο θεματολόγιο αυτό, πώς να το πω, μόνο για την επιβολή κυρώσεων σε αυτούς που δεν ε, προχωρούν, αλλά θέλουμε, παραλαμβάνω, να εμψυχώσουμε, να κινητοποιήσουμε όλους τους φορείς, να κινητοποιήσουμε τους ε, διοικητικούς κυβερνητικούς μηχανισμούς, αλλά και όλους τους άλλους φορείς. Είναι πάρα πολύ ευρύ το θεματολόγιο και άκρος πολύπλοκο. Δεν μπορεί λοιπόν να επιτευχθεί μόνο μέσω των κυβερνήσεων, απαιτεί συνεργασία και όλων των άλλων φορέων. Όταν είναι κανεί στι Βρυξέλλες, πολλές φορές έχει την εντύπωση ή ακούει ότι δεν γίνονται και πολλά. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Αντιθέτω, γίνονται πολλά. Λάβαμε αιτήσει από πάνω από 100 χώρες για τη στήριξη ελοποίηση των στόχων. Και αυτή τη στιγμή στέλνουμε και έχουμε ήδη στείλει σε πολλές χώρες αντιπροσωπείες αποστολές που περιλαμβάνουν μέλη διαφόρων ε, οργανώσεων ε, υπό την αιγίδα του UNDP, του Αναπτυξιακού Προγράμματος των ΗΕ. ΕΕ. Τους λέμε δηλαδή ποιο είναι το θεματολόγιο, ποιοι είναι οι στόχοι και βλέπουμε πού βρίσκονται. Είναι ευθυγραμμισμένοι στόχοι, υπάρχουν κενά, πού είναι αυτά τα κενά και πώς μπορούν να καλυφθούν γρήγορα. Ποια είναι η βάση αναφοράς, ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται, πολλά κινούνται εκεί έξω και αυτό ήθελα να το τονίσω για τη σημερινή μου παρουσίαση, ότι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πολύ σημαντικός, διότι όπως ακριβώς δεν είναι μόνο κυβερνητική ευθύνη, οφείλω να πω ότι και τα κοινοβούλια έχουν θεμελιώδη ευθύνη, πολύ σημαντική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων. Δηλαδή πρέπει να φροντίσουν η καλή θέληση της κυβέρνησης, γιατί οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων υπέγραψαν το θεματολόγιο και δεσμεύτηκαν γιατί παρότι θα χρειαστεί να σας πω ότι δεν είναι οι στόχοι του βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, αλλά των κρατών μελών. Όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πρόεδρε, πρωθυπουργοί υπέγραψαν. Δική του είναι ατζέντα, δικό τους είναι το θεματολόγιο και είμαστε όλοι εκεί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα Ηνωμένα Έθνη, οι εθνικές, ε, οι εθνικοί οργανισμοί ανάπτυξη και υποστηρίζουμε τους στόχους αυτού. και οι κυβερνήσει ή μάλλον καλύτερα οι χώρε είναι αυτέ που πρέπει να εφαρμόσουν. Ποιο είναι ο ρόλο τώρα των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι να αποκρισταλώσουν αυτού του στόχου σε συγκεκριμένε ενέργειε, να επιβλέπουν την επιτήρηση, να βλέπουν ότι συμμορφούνται με του στόχου, γίνεται σωστά εφαρμογή και παρακολουθούν ε, και τι έχει γίνει σχέση με τους ήδη εκτελεσθέντες στόχους. Πού πήγαν τα κονδύλια, πως διατέθηκαν ώστε η καλή βούληση να μεταφράζεται σε εφαρμογή και σε έργα, σε πράξεις. 15 χρόνια, φιλόδοξο το χρονοδιάγραμμα, υπάρχει αυτή η διαδικασία παρακολούθησης και όλοι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε στο χρονοδιάγραμμα αυτό και στις πολύ ισχυρές αυτές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί Πρέπει να πω ότι όταν ε, μιλώ με βουλευτέ όπω από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Επιτροπή Ανάπτυξη του Κοινοβουλίου, βλέπω ότι γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα. Δεν είμαι βέβαιο τόσο ότι υπάρχει το ίδιο επίπεδο γνώση και δέσμευση σε άλλε επιτροπέ. Και αυτή είναι μια πρόκληση για όλου μα. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ανάπτυξη. Πολύ ευρύτερο είναι πλέον το θεματολόγιο. Και αυτήν την έννοια θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες καλές εμπειρίες από διάφορες χώρες η Ουγγάντα, για παράδειγμα, δημιούργησε ένα κοινοβουλευτικό φόρουμ για τις στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι ε, εγκάρσιο, δηλαδή καλύπτει όλες τις επιτροπές και ενθαρρύνει το διάλογο και την ανάλυση, δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση και προσπαθεί να δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες. Το Τρινδάτ τον Πάγκο δημιούργησε μια ειδική επιτροπή για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη με ευθύνη συνολικά για το θεματολόγιο. Δηλαδή θα δουν τη χρήση της ενέργειας, του νερού, την εκπαίδευση, τη λογοδοσία των κυβερνήσεων, την κινητοποίηση των εθνικών πόρων και ούτω καθεξής. Αλλά και χώρες όπως το Πακιστάν έχουν μια task force για τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στην συνέλευση. Που σημαίνει ότι πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση. Δυστυχώς μέχρι τώρα κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο και νομίζω ότι μέρος της δικής σας ευθύνης από τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, τις Επιτροπές Ανάπτυξης, νομίζω ότι αν είχα να απευθύνω μια έκκληση σε εσά, θα ήταν να, να δείτε τι ε, σημασία έχει στις χώρες σας και στα κοινοβουλία σας και τι μπορείτε να κάνετε. Ήδη στη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προσπάθειες Υπάρχει ένα περιφερειακό νομοθετικό συμβούλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη που κάνει την παρακολούθηση, την παρέχει υποστήριξη και προωθεί το διάλογο. Και αυτά είναι καλά παραδείγματα από αυτά τα φόρουμ πολιτικής υψηλού επίπεδου, τα οποία μπορούν να βρουν μιμητές, πιστεύω. Τα Ηνωμένα Έθνη και συγκεκριμένα το πρόγραμμα ανάπτυξη στην προκειμένη περίπτωση έχει δημιουργήσει και ένα εγχειρίδιο και μια εργαλειοθήκη για τα κοινοβούλια. Συνεργαζόμαστε με πολλά κοινοβούλια ε, από τι διάφορε υπήρου. τι βοηθούμε να αξιολογήσουν τι δυνατότητε του, τι δεξιότητέ του, να μετρήσουν με τα εργαλεία που παρέχουμε ε, πώ τα πηγαίνουν στι διάφορε πολιτικέ και όποιοι ενδιαφέρεστε θα σα δώσουμε τα link, ε, του συνδέσει για το manual αυτό, το εγχειρίδιο αυτό και την εργαλειοθήκη δύο πολύ χρήσιμα εργαλεία κατά την άποψή μα. Εδώ θα σταματήσω εγώ. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι μέχρι τώρα. Δεν θα κάνουμε τα ίδια με το στόχο βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε να αλλάξουμε παράδειγμα. Δεν είναι βιώσιμη κοινωνία όσα έχει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι βιώσιμη για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, καταναλώνουμε, κινούμαστε στο περιβάλλον, ποιο είναι το οικονομικό μοντέλο, μεταφορές, δεν είναι βιώσιμος αυτός ο τρόπο διαβίωση και πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι την καθημερινότητά μα, τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Πρέπει να αλλάξουμε τις πολιτικές μας. Και αν θέλουμε να πετύχουμε θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι. Και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνεργαστεί με το δημόσιο τομέα. Αλλά και οι εταίροι πρέπει να ενθαρρυνθούν. Αυτή λοιπόν η συνέντευξη είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. αυτή η αντίληψη. Εταιρικέ σχέσει. Και ο 17ο στόχο συγκεκριμένα μιλά για συμπράξει, για εταιρικέ σχέσει. Δεν θα πάμε να πούμε τι πρέπει να κάνουν και να του δώσουμε απλά χρήματα. Είναι κάτι πιο ε, ευρύ, γιατί έχουμε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Υπάρχει και το θέμα το μεταναστευτικό. Εγώ δεν το λέω κρίση μεταναστευτική, αλλά μεταναστευτικό ζήτημα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις χώρες εταίρους που οδηγούν πολλούς στη φυγή από τις πατρίδες τους και να αναζητήσουν καλύτερο μέλλον εδώ στην Ευρώπη. Θέλουμε εκεί να τους εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στις χώρες τους. Θέλω να σας συγχαρώ που έχετε οργανώσει αυτή την μερίδα και να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την πρόσκληση. so Λοιπόν, η πρόκληση για μας είναι να βρούμε κοινέ λύσεις στα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον πλανήτη μας, που μοιραζόμαστε όλοι. Τα εθνικά κοινοβούλια σίγουρα έχουν ρόλο να διαδραματίσουν. Κάποιες από τις χώρες έχουν ήδη υποβάλει εκθέσεις στο υψηλό ε, πολιτικό στο φόρουμ υψηλού επίπεδου στα Ηνωμένα Έθνη. Φαντάζομαι θα είναι διαθέσιμε οι εκθέσει. Μπορείτε να τα δείτε διαδικτυακά. Δεν έχω τον κατάλογο μπροστά μου για τι χώρε που έχουν υποβάλει εκθέσει, αλλά πολλέ έχουν υποβάλει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει τον Ιούλιο του 2018. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας ε, τι κάνει το κοινοβούλιο σας ε, για να ε, λογοδοτούν τα κοινοβούλια για τις υποσχέσεις που έγιναν στη Νέα Υόρκη πριν από δύο χρόνια. Τώρα θα δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ελένη Θεοχάρου, η οποία θα προεδρεύσει στο πρώτο πάνελ για τη συνένεση για την ανάπτυξη, για να δούμε πώς θα προχωρήσει η εξωτερική ε, πολιτική για να επιτύχουμε τους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το λίκνο της δημοκρατίας όπως το θεωρούμε. Χαίρομαι που συντονίζω αυτή την ε, σημαντική συνεδρίαση. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπάρμπαρα για την εισαγωγή της και θα ήθελα να επαναλάβω το καλησέρισμα της Προέδρου μας στην αρχή της συνεδρίασης. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω και την εκτίμησή μου για την σημερινή σας παρουσία εδώ. Έχουμε μέλη του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, όπως αναφέρθηκε ήδη, από την Ισία, Νιγηρία, Μαρόκο και ε, φυσικά και εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων 25 χωρών Δεν ξέρω αν είναι όλοι εδώ, αλλά ε, να σας καλωσορίσω όλους. Ε, είμαι η Ελένη Θεοχάρους, ε, είμαι από την Κύπρο και είμαι μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε απάντηση στο θεματολόγιο του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες σημαντικές διεθνείς συμφωνίες οι οποίες εγκρίθηκαν επίσης το 2015, όπως για παράδειγμα η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, το πλαίσιο για την μείωση των ε, ε, ε κινδύνων και το ε, σύμφωνο της Αντίσα Αμπέμπα για την οικονομική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια αναθεώρηση της πολιτικής ανάπτυξης και συνεργασίας που καθορίστηκε βάσει και της συναντήληψης του 2005. Ο στόχος ήταν να υπάρχει ε, μία δέσμη μέτρων για να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να προσαρμοστούμε στις παγκόσμιες προκλήσεις όπως η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η ασφάλεια. Για μένα προσωπικά πρόκειται για κρίση, δεν αποτελεί απλώς ένα ζήτημα και εμείς από τον Ευρωπαϊκό Νότο το βιώνουμε ως κρίση. Όπω ε, πολύ σωστά λέει ο τίτλο αυτού του τμήματο τη συνεδρία, η Ευρωπαϊκή Συναντήληψη για την Ανάπτυξη αποτελεί την ευρωπαϊκή απάντηση στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη στι αναπτυσσόμενες χώρε. Η σημασία της νέας ευρωπαϊκής συναντήληψης ε, εδράζεται σε μια κοινή συνεκτική θέση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη για τους στόχους, τις αξίες, τις αρχές ε, και τις κύριες πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής και ε, συμπεριλαμβάνει φυσικά και την υλοποίησή της. Η Νέα Ευρωπαϊκή Συναντήληψη για την Ανάπτυξη υπεγράφει από κοινού από το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2017 και η Επιτροπή μας είναι αρμόδια για τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και κατάφερε να καταλήξει σε μια συμφωνία. Κατ' εξαίρεση ε, υπήρχαν δύο συνεισηγητές ε, ακριβώς για να εγγυηθούμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση ε, και ε, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συνεισηγητές, ε, ο αξιότιμος και έμπειρος συνάδελφος ο κύριος Βέντα και ο κύριος Νόιζερ, είναι εδώ μαζί μας σήμερα και θα σας δώσουν κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες οδήγησαν στην έγκριση της αντίληψης και στα βασικά χαρακτηριστικά της. Ο κύριος ε, Γκασπάρ Φροντίνη στη συνέχεια, ο Διευθυντής για τη Διεθνή Συνεργασία και Πολιτική Ανάπτυξη ε, στη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, ε, θα σας πει κάποια περισσότερα πράγματα για την εφαρμογή της συναντήληψης και το πώς εντάσσεται στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Τέλος, θα δώσουμε το λόγο σε όλα τα μέλη για να μιλήσουν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βέντα για τέσσερα λεπτά. με δικτάτορα εδώ που επιβάλλει τα χρονικά όρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσω θερμά όλους και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι Ακούστηκαν πολλά μέχρι τώρα. Η Ευρωπαϊκή Συναντήληψη για την Ανάπτυξη είναι μια κοινή ε, πολιτική δήλωση του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν χαρά για μένα να εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των οποίων ηγήθηκε η Μαλτέζικη Προεδρία. Μαζί με τους συναδέλφους ε, ε, και με την υποστήριξη της Προέδρου μας καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία προκειμένου ε, να ε, καταλήξουμε σε αυτή τη συνένεση. Γιατί χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση λοιπόν στην αναπτυξιακή πολιτική. Το ανέφεραν και οι προλαλήσαντες. Όταν εξετάζουμε την πολιτική κατάσταση, τη διεθνή κατάσταση, υπάρχουν νέες προκλήσεις Οχτώ στόχοι της χιλιετέας ε, έχουν περάσει και έχουν μεταφραστεί σε 17 βιώσιμους στόχους ανάπτυξης και επομένως χρειαζόταν μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση, μια νέα ε, συναντήληψη η οποία θα συνδυάζεται με το θεματολόγιο του 2030 και τους στόχους του. Ε, επομένως ένα ευρύτερο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα επικεντρώνεται στους ανθρώπους, ε, στην ειρήνη, στην ευημερία, στην εταιρική σχέση. Επομένως, ε, η συναντήληψη αυτή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, διότι αλλάζει το πλαίσιο της συνεργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθορίζει νέες προτεραιότητες όσον αφορά τη μείωση της ένδυας, τη βιώσιμη ανάπτυξη βεβαίως, την ε, εξάλληψη των ανισοτήτων και πολλές άλλες προκλήσεις οι οποίες ε, αφορούν δημογραφικές αλλαγές, οικονομικές αλλαγές, κοινωνικά προβλήματα και περιβαλλοντικά προβλήματα. Όπως ε, όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι από τους μεγαλύτερους χορηγούς, δίνουν τα μεγαλύτερα κονδύλια, 77,5 ε, εκατομμύρια για εκπαίδευση, καλή διακυβέρνηση, κράτος δικαίου, πρόσβαση στην υγεία, ισότητα των φύλων, πρόσβαση σε νερό και πρώτες ύλε, καθώς επίσης και δημιουργία θέσεων εργασίας ε, και καινοτομία. Η άλλη πλευρά του νομίσματος βέβαια είναι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία αποτελεί και το θεμέλιο της συναντήληψης και της δέσμευσή μας ε, για ε, χρηματοδότηση. Το 0,7% του ΑΕΠ για αυτό το συγκεκριμένο στόχο μέχρι το 2030. Από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ σημαντικό η συνένεση, ε, η συναντήληψη να αναφέρει ε, τη συνέπεια και ε, όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τη χρηστή διακυβέρνηση τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να υπάρχει λογοδοσία και δέσμευση. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο, ο, να ενισχύσουμε και το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς επίσης και τις τοπικές, περιφερειακές κυβερνήσεις και την ίδια την κοινωνία των πολιτών. Και εδώ αναφερόμαστε σε πολιτική υποστήριξη, σε στήριξη στον προπολογισμό και δημοκρατική ε, εποπτεία, δημοκρατικό έλεγχο στις χώρες μας, αλλά και σε άλλες χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες για παράδειγμα η μεγαλύτερη δέσμευσή μας και οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα που αφορούν ε, το ισότιμο δίκαιο εμπόριο, αποτελεί ε, πολύ σημαντικό μοχλό αυτής της συναντήληψης. Όλα αυτά συνδυάζονται με την ασφάλεια ε, και την κατάλληλη πολιτική μετανάστευσης, διότι αν εξετάσουμε όλες αυτές τις κρίσεις διαπιστώνουμε ότι αποτελεί ένα πόσπαστο τμήμα της ε, λύσης. Η καταπολέμηση της, εξαναγκαστικής, της καταναγκαστικής ε, μετανάστευσης ε, είναι στη ρίζα του προβλήματος. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Αν υπάρξει λοιπόν κατάλληλη πολιτική ασφαλείας, πολιτική σε οικονομικά θέματα, περιβαλλοντική πολιτική, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε καλύτερη διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι με αυτά μπορώ να ολοκληρώσω και να δώσω λίγο το λόγο στον Όρμπερντ. Παρακαλώ. Okay, thank you very much. Uh, Eleni. Ευχαριστώ πολύ Ελένη. Ευχαριστώ πολύ Μπόγκταν. Αγαπητοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, από τα Αφρικανικά Κοινοβούλια και το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό σημάδι εν ώψη και τη επικείμενη διάσκεψη κορυφή μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρικανικών χωρών, που είστε εδώ σήμερα για να συζητήσετε μαζί μα την υλοποίηση και τι δυνατότητε ε, που προσφέρουν οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη. Εγώ σα ομιλώ ω συνεισηγητή από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για το θέμα, το οποίο συνδιαπραγματεύθηκα με τον Μπόγκταν Βέντα, το συναλφό μου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μια παρατήρηση. Είμαι Γερμανό και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συνένεση κοινή αντίληψη, αν θέλετε, στη Γερμανία σε ό,τι αφορά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Ωστόσο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταφέραμε να έχουμε συνένεση για τη συνένεση, για την κοινή αντίληψη που σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και δεν μιλώ μόνο για τις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες αλλά και για τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου. Οι συνάδελφοί μου και εγώ προσωπικά θεωρούμε ότι η εκρίζωση της στόχιας ε, παραμένει ο παρεξάρχων στόχος, πρωταρχικός στόχος της κοινή αντίληψης. Το ίδιο και μια συνεκτική αναπτυξιακή πολιτική. Η εκρίζωση της ε, σημαίνει ότι πρέπει οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική διάσταση να ληφθεί υπόψη και να ευθυγραμμιστεί ε, για, με τους στόχους 2030. Ε, και για την επίτευξη των στόχων αυτό θα πρέπει τα κράτη-μέλη να πετύχουν ε, το στόχο του 0,7 τη επίσημη ανεπτυξιακή βοήθεια. Είναι κάτι για το οποίο πιέζουμε στι διαπραγματεύσει και η κοινή αντίληψη μέχρι στιγμή δεν έχει ένα νέο χρονοδιάγραμμα για ενδιάμεσου στόχου. Κάτι το οποίο ε, είχαμε πει στην προηγούμενη κοινή αντίληψη. Γι' αυτό λοιπόν βασιζόμαστε σε εσά να επιμείνετε να πετύχουν τα κράτη-μέλη σας στο στόχο του 0,7. Σε ό,τι αφορά τώρα την κλιματική αλλαγή, και αυτή είναι σαφής προτεραιότητα, είναι κοινή αντίληψη, επανεπιβεβαιώνει τις δεσμεύσεις της COP21. Η κλιματική αλλαγή έχει στενή σχέση με τη γεωργία, ε, την σκαλλιέργειες ε, για να καταπολεμήσουμε και τον υποσυτισμό και τη φτώχεια θα πρέπει επενδύσει να υποστηρίξουν τους γεωργούς με τους κατάλληλα προσαρμοσμένους μηχανισμούς. Θα πρέπει να στηρίξουν τις γεωργοεπιχειρήσεις ε, και τους συνεταιρισμούς. Στενά συνδεδεμένες με τις επένδυσεις και το εμπόριο είναι οι κοινωνικές περιβελιακές πτυχές και τα σχετικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται λοιπόν σε αυτή την κοινή αντίληψη κίνητρα ώστε να ενταχθεί η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε αυτές τις προσπάθειες και να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα για επενδύσεις τι όμενε χώρε. Εμείς οι βουλευτές πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να επιμείνουμε και να συνεχίσουμε να ε, παρακολουθούμε την εφαρμογή αυτών των προτύπων για να δούμε πραγματικές αλλαγές ε, στις συνθήκες διαβίωσης ε, των συμπολιτών. Για την ανθρωπιστική βοήθεια με παρατήσει επειδή δεν καλύπτεται στην κοινή αντίληψη. Είναι κάτι νομίζω που πρέπει να μας ασχολήσει περισσότερο. Βέβαια, εμείς στην Επιτροπή Ανάπτυξης ε, είμαστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι σε αυτή τη διάσταση. Βελτίωση της οδικών διαβίωσης θα περιορίσει τη μετανάστευση μακροπρόθεσμα. Η μετανάστευση βέβαια έχει και θετική συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη. Και η αντίληψη ζητά μια μεταναστευτική πολιτική που θα βασίζεται σε αμοιβαία λογοδοσία, σε πλήρη σεβασμό των υποχρεώσεων απέναντι ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα δεσμεύει τα κράτη-μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια δομημένη ολιστική προσέγγιση και για την αντιμετώπιση των ε, βασικών αιτιών της μετανάστευσης. Αναπτυξιακή βοήθεια και διαχείριση μετανάστευσης. Πλέον αυτή η διασύνδεση δεν έχει αρνητικές αποχρώσεις, χάρη στις προσπάθειές μας. Περιμένω και του χρόνου τον Νοέμβριο να σας ακούσω Πρώτα απ' όλα βέβαια τώρα για να δω τι γίνεται με την επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης της χώρας σας. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας καλωσορίσω και στην γλυκύτατη ελληνική γλώσσα. And uh, before I give the floor to Mr. Frondini, I will ask uh, our colleagues from the European Parliament if they want to take the floor to indicate it. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν επιθυμούν να λάβουν το λόγο να σηκώσουν το χέρι τους τώρα ή διαφορετικά οι ε, εκπρόσωποι των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων να συμπληρώσουν τις κάρτες που βρίσκονται στο έδρανό τους αν δεν τον έχουν ήδη κάνει αυτό. Κύριε Φροντίνη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Είμαι και εγώ ιδιαίτερα ευτυχή που έχω τη δυνατότητα να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο, σε εσά, για το ζήτημα τη κοινή αντίληψη για πολλού λόγου. αλλά ε, ιδιαίτερα επειδή η επίτευξη αυτή τη κοινή αντίληψη ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, αποτέλεσμα της καλής συνεργασίας που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και είχα ως, ε, από την πλευρά της Επιτροπής ε, και εγώ ως πρόσωπος της Επιτροπής μια πολύ καλή συνεργασία με ε, τους ε, εισηγητές. Θα περάσω αμέσω στην παρουσίαση γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Το πρώτο στοιχείο που θέλω και εγώ να τονίσω, που ήδη αναφέρθηκε, είναι ότι η κοινή αντίληψη έχει ε, την υπογραφή και την υποστήριξη στο υψηλότερο δυνατό ε, επίπεδο. Στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνοβουλίου και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διεξάγει την αναπτυξιακή της πολιτική, αλλά επίσης ε, δίνει και πολιτικές κατευθύνσεις, δίνει ένα πλαίσιο πολιτικής για τις διμερείς σχέσεις αναπτυξιακής συνεργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από την αναπτυξιακή πολιτική που κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και 28 διαφορετικές εθνικές αναπτυξιακέ πολιτικέ. Και πρέπει να ενισχύσουμε την συνοχή μεταξύ αυτών των 29 πολιτικών. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική ε, αναπτυξιακή πολιτική. Και η βάση για αυτήν την ε, προσπάθεια να αυξήσουμε τη συνοχή είναι το έγγραφο αυτό, η κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Σε αυτή τη νέα συναντήληψη προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων και να την προσαρμόσουμε στις αλλαγές στο διεθνές θεματολόγιο. Ακούστηκε ήδη πως αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο να αντιμετωπίζουμε την ε, διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία και γενικότερα τη διεθνή συνεργασία. Για το ζήτημα, για παράδειγμα, των προσφύγων μάλλον συγγνώμη, με το προηγούμενο σύστημα. Είχαμε στόχους για τις αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναπτυγμένες χώρες βοηθούσαν. Ε, ως αν οι αναπτυγμένες χώρες να μην είχαν προβλήματα. Ε, αυτό συνέβαινε με το παλιό σύστημα των στόχων της χιλιετίας. Με το νέο σύστημα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης προσπαθούμε να έχουμε συντονισμένη δράση και στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό αυτή τη νέα προσέγγιση προσπαθήσαμε να την αντικατοπτρίσουμε και στο ε, στη νέο ευρωπαϊκό κονσένσους. Μέσα από κάποιους, κάποιους πυλώνες, ε, την ευημερία, τους ε, πολίτες, το περιβάλλον, την ειρήνη. Και το τη διατυπώσαμε έτσι την πολιτική μας αυτή γιατί θεωρούμε ότι η αναπτυξιακή συνεργασία δεν μπορεί να ε, την εξετάζει κανείς ή να την εφαρμόζει ξεχωριστά από τις υπόλοιπες πολιτικές. Προσπαθούμε λοιπόν να εστιάσουμε στις σχέσεις που έχει η αναπτυξιακή συνεργασία με άλλες σημαντικές πολιτικές. Για παράδειγμα, με το ζήτημα της ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ειρήνη η μετανάστευση, είτε την ονομάσει κανείς κρίση, είτε πρόβλημα, είτε ευκαιρία, είναι ένα θέμα πάντως πολύ σημαντικό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα της ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, η οποία και αυτή πρέπει να συνδέεται, να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αναπτυξιακή συνεργασία. Επίσης υπάρχουν ε, σχέσεις με τις πολιτικές μας για την κλιματική αλλαγή, με τις, για την εμπορική συνεργασία, με την φορολογική πολιτική ξέρω δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ πειγραμματικά και στο πώς προσπαθούμε να, τα υλοποιήσουμε όλα αυτά. Όπως είπα, το πρώτο και σημαντικότερο είναι η βελτίωση του συντονισμού της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και των κρατών μελών αφετέρου. Γι' αυτό εξάλλου έχουμε και στη σημερινή συνάντηση εκπροσώπους και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούμε να βελτιώσουμε την συνεργασία, τον συντονισμό. Ε, και αυτό ε, συνεχίζεται και με τα διάφορα προγράμματα που εφαρμόζουμε επί τόπου. Δεύτερο είναι να δούμε τη χρηματοδότηση. Υπάρχει η ξεκάθαρη δέσμευση ότι θα πηγαίνει το 0,7% του ΑΕΠ των αναπτυγμένων κρατών για την αναπτυξιακή συνεργασία ή το 0,4% για την ανάπτυξη από τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά επίσης θα πρέπει να βρούμε τρόπους για να ε, εθνικών πόρων. Γιατί αυτή η πηγή χρηματοδότησης, η εθνική, πόρη, είναι η πιο σταθερή. Χρειάζεται επίσης να δούμε ε, την συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων μωρών πέραν από τις κυβερνήσεις και πέραν από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ε, γιατί αυτοί οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης αφορούν τους πάντες. Και γι' αυτό ε, πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία συζήτηση με εσά που εκπροσωπείτε τους λαούς των χωρών σας. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των διαφόρων πολιτικών. Επίσης υπάρχει το θέμα της συνοχής. Γιατί το σημαντικότερο πέρα από την εξέβριση χρημάτων είναι να έχει κανείς το σωστό μείγμα πολιτικής. Δηλαδή πολιτικές αναπτυξιακές συνεργασίε, οι οποίες να είναι συνεκτικές με τις υπόλοιπε πολιτικές. Και έτσι ώστε τελικά να βοηθούμε τις χώρες αυτές. Τέλος. Παρά γεγονό ότι η κοινή αντιλήψη εστιάζει στους στοχούς, στους στοχότερους, στην εξάλληψη της φτώχειας, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να προσαρμόζουμε την αναπτυξιακή μας συνεργασία στις διαφορές που υπάρχουν ε, ανάμεσα στις διάφορα κράτη του κόσμου. Ε, κάποιες χώρες βγαίνουν από μια κρίση, κάποιες χώρες βγαίνουν από έναν πόλεμο, κάποιες άλλες είναι ήδη σε μια τροχιά ανάπτυξης. Ε, αυτό είναι στοιχείο κλειδί για να να επιτύχουμε τους στόχους μέχρι το 2030, δηλαδή το να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα στοιχεία πολιτικής στην ενδιάμεση ε, αναθεώρηση που κάνουμε στο πλαίσιο του τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και να προετοιμαστούμε για το επόμενο ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πέραν αυτού, ε, αυτών έχουμε ξεκινήσει και συγκεκριμένες δράσεις το ευρωπαϊκό ε, σχέδιο επενδύσεων ε, στο οποίο προσπαθούμε να, με το οποίο προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις επενδύσεις στην Αφρική. Η συνεργασία με, το, με την UN Women, με το πρόγραμμα του ΕΕ για τις γυναίκες, για την αντιμετώπιση των διακρίσεων με βάση το φύλλο. Οι προσπάθειες που κάνουμε για την εξέβρεση εθνικών πόρων. Αυτά είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να δούμε και πώς κάθε χώρα, κάθε εθνικό κοινοβούλιο προσπαθεί να συμμετάσχει σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Κλείνω λέγοντας ότι ένας τρόπος για να έχουμε καλύτερη εφαρμογή της πολιτικής είναι να έχουμε καλύτερη παρακολούθηση της, δηλαδή αναφορές να δείχνουν πώς τελικά συνεισφέρει ο καθένας σε αυτούς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θα προετοιμάσουμε μια τέτοια έκθεση για το 2019 όταν θα γίνει η συνάντηση του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου. Θα ήταν, θα εκείνη τη στιγμή ένα κρίσιμο σημείο και θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε με την έκθεση αυτή τις πρωτοβουλίες που θα έχουν αναλυφθεί σε επίπεδο κρατών μελών και ένωση συνολικά. Ευχαριστώ κύριε Φροντίνη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε το λόγο τώρα. Θα έχετε τρία λεπτά ο καθένας. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να είστε συγκεκριμένοι για να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σε όλους. Σας παρακαλώ όταν παίρνετε το λόγο να μας συστήνεστε και να μας λέτε και από ποια χώρα είστε και αν ε, έχετε ερώτηση, σας παρακαλώ να μας πείτε ε, σε ποιον απευθύνετε την ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ξεκινούμε με την Άννα Τερών από την Ισπανία. Ε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνεδρίαση. Αυτή τη στιγμή λέγομαι Άννα Τερών από την Ισπανία. Μ' ακούτε? Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Εντάξει. Άννα Μπελέντερον από την Ισπανία. Και σήμερα το πρωί θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Δεν απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένα. Ε, είναι γενική ερώτηση προς το πάνελ όσον αφορά την κοινή αντίληψη. Διάβασα και κάποια πράγματα για το θέμα αυτό, για την διαδικασία αυτής της κοινή αντίληψης. Ε, διάβασα ότι ε, υπήρξε και κάποια εναλλεκτική κίνηση. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ε, τι στήριξη είχε αυτή η κοινή αντίληψη στο Κοινοβούλιο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μου διευκρινίσει αυτή την αμφιβολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άννα. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Άνικιν Βουίτφελτ από την Νορβηγία. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. So, thank you so much. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πολύ και για την ε, πρόσκληση σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Η ίση κατανομή πλούτου είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Η φορολογική παράδοση και οι διαρροές κεφαλαίων δυσχεραίνουν την εφαρμογή των προγραμμάτων παιδείας, τα νοσοκομεία και της πρόνοιας των χωρών. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κατάλληλη ηγεσία στις χώρες όσον αφορά την ίση κατανομή μεταξύ αλλά και εντός ε, των αναπτυσσόμενων χωρών. Και πιστεύω ότι η διεθνής βοήθεια μπορεί να διατηρηθεί μόνο αν οι πολιτικοί ηγέτες είναι υπόλογη για την αναδιανομή του πλούτου και την ε, ε, κατάλληλη ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη είναι κομβικός παράχων... και χαίρομαι ότι διότι τώρα Υπάρχει συγκεκριμένη αναπτυξιακή βοήθεια, περίπου 1% του ΑΕΠ, επειδή ακριβώς αποφασίστηκαν όλα αυτά και τα προώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ευρωπαϊκή Ευρώπη μάλλον αναπτύχθηκε λόγω του εμπορίου αλλά και της αναπτυξιακής βοήθειας και φυσικά ε, το άνοιγμα των αγορών ήταν σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη στη στρατηγική τους. Και πολλές χώρες ε, επιτυγχάνουν ανάπτυξη μέσω εμπορίου, αυξάνεται ο ανταγωνισμός από τις αναπτυσσόμενες χώρες όμως και αυτό οδήγησε σε αποφάσεις ελευθέρου εμπορίου και στεναρές αντιστάσεις σε πάρα πολλές χώρες ε, σήμερα και από την πολιτική αριστερά αλλά και από τη δεξιά εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού στην Ευρώπη, ε, θα υπάρχει προστατευτισμός. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Ο διεθνής ανταγωνισμός ε, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κατάλληλες θέσεις εργασίας. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ε, και να τον μετράμε, να γίνεται μέτρηση πολύ προσεκτικά για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Uh, ο κύριος Εμμανουελίδης από την Ελλάδα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη, ένα νέο πλαίσιο για μια κοινή προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική, που πρέπει να εφαρμόσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και τα κράτη-μέλη της στη συνεργασία τους με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνειδητοποιούμε ότι για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Την ανεργία των νέων, τις αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών και την προσφυγιά, την κλιματική αλλαγή και τη θέρμαση του πλανήτη, τη φτώχεια αλλά και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι συχνό φαινόμενο σε πολλά σημεία του πλανήτη. Η εφαρμογή της Ατζέντα 2030 μπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων αυτών. Σε εθνικό επίπεδο, συντονιστικό ρόλο για την ενεργοποίηση των ε, εμπλεκομένων θεματικά Υπουργείων ανέλαβε από το Δεκέμβριο του 2016 η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης παράλληλα με το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να ενσωματωθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής. Σε πρώτη φάση, οι 17 στόχοι και οι 169 υποστόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η χώρα μας ενσωματώνονται και ισορροπούν με τις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική οι οποίες άλλωστε τρεις αυτές διαστάσεις αποτελούν τις βασικότερες προϋποθέσεις για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για την ανθρωπότητα. Εκείνο που θα πρέπει όλοι στο βαθμό που μας αναλογεί να φροντίσουμε είναι ε, αυτές οι διακηρύξεις να περάσουν σε ένα στάδιο υλοποίησης γραφής σε αυτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Μανουή. Now we give the floor to Mrs. Rosalia Biro, Biro. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Ροζαλία Μπυρό από τη Ρουμανία. Εδώ είμαι. Πρώτα απ' όλα, να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση τη σημερινή συνάντηση. Είναι πολύ σημαντική για εμάς. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω λιγάκι την ε, κατάσταση ε, στη Ρουμανία και θα μιλήσω στα ρουμανικά. Η Ρουμανία είναι ένα κράτος από το 193 του ΙΕ που από το 2015 υποστηρίζει τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και το, ε, η κυβέρνησή μας έχει προσπαθήσει να καταρτήσει ένα εθνικό ε, σχέδιο υλοποίησης των στόχων αυτών με βάση την προσπάθειά μας να καταλήξουμε σε μια κοινωνία στην οποία θα καταπολεμηθούν οι αποκλεισμοί και οι διακρίσεις. Εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να βρούμε ποιοι είναι οι μηχανισμοί που θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε αυτούς τους στόχους, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί να σταματάνε ε, την υλοποίησή τους, να έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης τους και ε, να βρούμε ε, τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μια ενιαία προσέγγιση στο κοινωνικά, στα οικονομικά θέματα και στα ζητήματα του περιβάλλοντος αντιμετώπιση αυτών των τριών ε, πτυχών από κοινού. Επίσης, πιστεύω ότι το πρώτο στάδιο ε, που χρειάζεται είναι να κάνουμε μια χαρτογράφηση των εθνικών στρατηγικών για τα διάφορα θέματα που καλύπτονται από τους στόχους ε, βιώσιμη ανάπτυξης. Δηλαδή, την πολιτική για το περιβάλλον, την πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων και την πολιτική για την αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτε χώρες. Μετά θα πρέπει να δούμε στις εθνικές αυτές στρατηγικές, αυτέ τι εθνικές πολιτικές που υπάρχουν κενά. Και μετά να καταλήξουμε σε μια στρατηγική με προθεσμίες ε, και με ξεκάθαρες αρμοδιότητε Δημιουργήσαμε ένα ε, ξεχωριστό ε, μια ξεχωριστή γραμματεία υπό την ευθύνη του Πρωθυπουργού, που λογοδοτεί στον Πρωθυπουργό, η οποία έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και το θεματολόγιο 2030 στην ε, Ρουμανία. Αυτή τη στιγμή το Ρουμανικό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαβούλευση την οποία προσπαθούμε να συμμετάσχουν εκπρόσωποι και από τη δημόσια διοίκηση ε, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχει επίσης δημιουργηθεί ε, ένα διυπουργικό συμβούλιο μέσω του οποίου προσπαθούμε να συντονίσουμε τις στρατηγικές που έχουν οποιαδήποτε ε, επίπτωση στο περιβάλλον. Και το Υπουργείο Περιβάλλοντος ε, συμμετέχει στην κατάρτιση των εθνικών στόχων. Επίσης, η Επιτροπή Εξωτερικών του Ρουμανικού Κοινοβουλίου προσπαθεί να ενθαρρύνει και να προωθήσει την ε, εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Προσπαθούμε να γίνουμε κόμβος ε, στην προσπάθεια υλοποίησης αυτών των στόχων στην Ανατολική και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Και, προετοιμαζόμαστε επίσης και για τη δημιουργία 2018. Σας ευχαριστώ. Thank you, uh, Πριν να δώσω τώρα το λόγο σε δύο συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, την κυρία Λόλα Σάντσες και την κυρία ε, Χάιντι Χάουταλα, θα ήθελα να απαντήσω, αν θέλετε, στην κυρία Τερών, στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Τερών. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην Ολομέλεια ήταν 405 βουλευτές υπέρ, 70 κατά και 159 αποχές στο ψηφοφορία για την κοινή αντίληψη. Λόλα. Ευχαριστώ, Ελένη η επικαιροποίηση της κοινή αντίληψης θα έπρεπε να χρησιμεύσει για να ευνοήσουμε τη λογική των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης ε, και των πολιτικών, θέματα στα οποία έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά τελικά χρησιμοποιήθηκε για να δεσμεύσουμε τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την ανάπτυξη και να θεμελιώσουμε το ρόλο του ιδιωτικού τομέα. Ε, ουσιαστικά χρησιμοποιείται επίσημα η ανάπτυξη για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών, που σημαίνει ότι εξωτερικοποιούμε τον έλεγχο των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες χώρες. Θέλουμε να ενισχύσουμε μηχανισμούς με τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει το blending και η συμπράξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, χωρίς να λάβουμε υπόψη μας τις λογικές αμφιβολίες που προκύπτουν. Δεν λαμβάνεται υπόψη και το θέμα της υποχρεωτικής ευθύνης του ιδιωτικού τομέα σε θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θέματα που αφορούν ε, το φύλλο είναι πολύ αποδυναμωμένα, ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τους ε, ΛΟΑΔ και δεν λαμβάνεται καμία ε, μέρημνα για την παρακολούθηση της προόδου για την κοινή αυτή αντίληψη. Είναι παράδοξο λοιπόν να θεωρείται κοινή αντίληψη όταν το ψήφισε το 54% του Κοινοβουλίου οι φιλελεύθεροι, το EFTD, η πράσινοι και η ε, ενωτική αριστερά προτείναμε ένα εναλλακτικό ψήφισμα στο οποίο ε, αναφερόμασταν και στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πολύ απέχει από το τελικό κείμενο επαναλάβαμε ότι πρέπει να έχουμε τις αρχές της αποτελεσματικότητας, τη βοήθεια για την ανάπτυξη, ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές των χωρών εταίρων, τη διαφάνεια και επίσης τη λογοδοσία όλων των εμπλεκομένων ε, φορέων στην ε, διαδικασία. Και επίσης ε, θέλαμε να έχουμε μηχανισμούς λογοδοσίας για να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ. Και επίσης προσπαθούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να ε, επιτευθούν σταδιακά αυτοί οι στόχοι. Επαναλάβουμε ότι η βοήθεια για την ανάπτυξη δεν πρέπει να γίνεται υπό όρους για τη συνεργασία των χωρών που λαμβάνουν την ενίσχυση για θέματα μετανάστευσης και ασφάλειας και απορρίψαμε οποιαδήποτε προσπάθεια να ε, ε, σχετιστεί βοήθεια με τον έλεγχο των συνόρων και τις υποχρεωτικές επιστροφές. Και τέλος επισημάναμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μας αυστηρά την πρόσφατη μεταρρύθμιση της βοήθειας για την ανάπτυξη για να χρησιμοποιούνται μέσα για την ανάπτυξη στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας και να τα σχετίσουμε με τον σαφή στόχο της εκρίζωσης της ένδυας και της θεμελίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι η κοινή αυτή αντίληψη είναι πολύ αδύναμη για μια πολύ αδύναμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Λόλα. Θέλετε τώρα το λόγο. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω και μπορώ να απαντήσω και ισπανικά. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν μόνο 55% στο Λομέλια, γιατί 77,8% ήταν το ποσοστό αυτό υπέρ της συνένεσης. 10% ήταν κατά και κάνα 12% περίπου απήχαν από την ψηφοφορία. Που σημαίνει ότι σχεδόν το 80% ψήφισε υπέρ της συνένεσης. Άρα μην δίνετε στοιχεία τα οποία δεν είναι αληθή. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ξέρετε πολύ καλά ότι διαπραγματευτήκαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις πολιτικές ομάδες. Φυσικά και υπάρχουν κάποιες πτυχές που σε ό,τι αφορά την ομάδα που εκπροσωπείς εσύ ήθελα ε, να, εστιάσουμε αλλού σε σχέση με εκεί που εστιάζα. Αλλά το θέμα είναι να βρεθεί ένα συμβιβασμός. Μη λέμε όμως πράγματα που δεν ισχύουν ότι τότε στην Ολομέλεια ότι ήταν 693 βουλευτές, εκ των οποίων οι 77,8 ψήφισαν υπέρ και να αλλάζουμε τώρα τα στοιχεία. I will give the floor uh, later to... Θα δώσω αργότερα το λόγο στην Heidi, γιατί θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον κύριο Μαμέτη Σιντίπεμ από το Παναφρικανικό, Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Merci, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πρόγραμμα μας ζητήθηκε να λάβουμε και εμείς το λόγο. Και το θέμα μας είναι η συνένεση, που ουσιαστικά είναι μια ευρωπαϊκή συνένεση, μια ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη. Πιστεύω όμως πως σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να υπάρχει μια πλανητική συνένεση σε όλες τις ε, πιθανές υποθέσεις και σενάρια. Αυτή η ευρωπαϊκή συνένεση θα πρέπει να προσεγγίσει, αν θέλετε, την Αφρικανική συνένεση λόγω και της κοινή μας ιστορίας. Γλωσσικής, γιατί εγώ όπως ακούτε μιλάω γαλλικά, και βέβαια έχουμε και πολιτικές, οικονομικές και ανθρώπινες σχέσεις μακραίωνες. Χθες ακούσαμε να λέγεται το Πάπο ότι έχει αναπτυχθεί η Ευρώπη αλλά και με τη συμβολή ε, της Αφρικής. Εμείς θέλουμε να βασιζόμαστε ως Αφρική και στους εαυτούς μας αλλά και στην ιστορική σύμπραξη, στην ιστορική εταιρική σχέση με την Ευρώπη. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης όμως, θα πρέπει να έχουμε ενήλικες σχέσεις ε, Δηλαδή ο ένας αντιμετωπίζει τον άλλο ως ενήλικο. Υπάρχει και ένας ε, στόχος πολύ σημαντικός για την Αφρική, ο υπαριθμών 17. Αλλά όλοι οι στόχοι είναι προτεραιότητες. Και πάρα πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να δούμε πού υπάρχει σύγκληση συμφερόντων. Η ανάπτυξη της Αφρικής, κατά τη δική μας άποψη, θα περάσει από τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Υπάρχουν προκλήσεις λόγω της κλιματικής απορρίθμισης. Το είπε και ο πρόεδρος. για το τσάντ και τις δραστηριότητες που υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φεύγουν. Γιατί φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κάπου που είναι καλύτερα. για την ε, απεικιοποίηση, απεικιοκρατία, για ε, τα προβλήματα που υπήρχαν. Για, τις, για τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Χρειάζεται μια πλανητική αντίδραση για την επίτευξη των στόχων. Οι 17 στόχοι σε ό,τι αφορά την, τον προγραμματισμό, αν θέλετε, για τις χώρες μας και για τη δεκαετία αυτή. Είχαμε και το θεματολόγιο του 2030, αλλά είχαμε και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αν είναι λίγοι μαθητές σε μια τάξη όμως, πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Χρειάζονται εσωτερικέ προσπάθειες, σίγουρα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είναι μοιρασμένε οι προσπάθειες για να υπάρχει και μοιρασμένη ανάπτυξη και στην Αφρική, που βέβαια αυτό θα ωφελήσει και την Ευρώπη. Υπάρχουν οικονομικοί πόροι η Αφρική χρειάζεται την ανάπτυξη. Το μέρισμα, αν θέλετε, μπορεί να μας ωφελήσει όλους. Κύριε Μαμέτη, με συγχωρείτε, λέει πρόεδρος, αλλά οφείλω να σας διακόψω. Έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω εδώ αυτό που είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα. Για να πετύχουμε την ανάπτυξη πρέπει να επενδύσουμε στην παιδεία, στην παιδεία και πάλι στην παιδεία. Αυτό ήταν το βασικό δόγμα και είναι και εδώ το βασικό δόγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκ Έντζελ από το Λουξεμβούργο. Και παρακαλώ όλες και όλους τους ομιλητές να τηρείτε το χρόνο των τριών λεπτών. Διότι αλλιώς θα πρέπει να διακόψουμε και δεν θα έχετε λάβει όλο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε ό,τι αφορά τη συνένεση για την ανάπτυξη. Από πλευρά Λουξεμβούργου δεν θεωρούμε ότι πρόκειται για πρόοδο, αλλά για πιστοδρόμηση σε σχέση με την προηγούμενη συνένωση του 2005. Βέβαια, το καλό είναι ότι έχει ευθυγραμμιστεί με το θεματολόγιο 2030 και του 17 στόχου βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο είναι συνεκτικό. Προσπαθεί δηλαδή ε, να κάνει πιο ε, συνεκτικές μεταξύ τους τις διαφορετικές αναπτυξιακές πολιτικές των 27. Όμως, νομίζουμε ότι έχει παρεκκλίνει από τη βασική αρχή που ήταν η κρίζωση της φτώχειας αυτή η νέα συνένεση. Το δεύτερο που μας ανησυχεί και ο υπουργό μα το εξέφρασε, εξέφρασε τι ανησυχίε του πολλέ φορέ ε, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ότι οι όροι και προποθέσει, ε, η αναφορά σε συμφωνίε επανεισδοχή ε, είναι κάτι που δεν μα ικανοποιεί. Επίση, σε ό,τι αφορά ε, τα κριτήρια της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΣΑ για την πρόσβαση στην ανάπτυξη και την ασφάλεια. Και αυτά κάπως μας ανησυχούν, γιατί έχουν συμπεριληφθεί στη συνέντευξη. Και όπως είπε και ο κύριος Νόιζα, ο Γερμανός ε, βουλευτής, δεν υπάρχει σύστημα παρακολούθηση ή χρονοδιάγραμμα για την παρακολούθηση της επιτέξης του στόχου του 0,7%. Πράγματι αυτό λείπει από τη νέα συνένεση και είναι κρίμα. Αυτά ως παρατηρήσει σε σχέση με τη συνέντευξη. Μια άλλη παρατήρηση τώρα, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μοντέρο από τα Ηνωμένα Έθνη για τη σημασία των ε, κοινοβουλίων και του ρόλου τους. Πράγματι είναι μεγάλη σημασία των Εθνικών Κοινοβουλίων για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, Όχι όμω μόνο ω αλληλεπίδραση με τι κυβερνήσει, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε στο Λουξεμβούργο μια Επιτροπή ανάπτυξης, που οργανώνει πολύ τακτικά και τι έχει θεσμοθετήσει ανταλλαγέ με βουλευτέ και μέλη τη κοινωνία των πολιτών, κυρίω ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης, ε, της ανάπτυξης. Νομίζω ότι και αυτή η δραστηριότητα είναι σημαντική. Το Λουξεμβούργο πρέπει να πω ότι ε, έστειλε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου μαζί με ε, την κυβέρνηση στις ΗΠΑ, ε, στη Νέα Υόρκη. Και είχαμε ήδη ενημερωθεί για το τι θα συζητεί το εκεί και όταν επέστρεψαν μας ενημέρωσαν εκ νέου για το τι συζητήθηκε. Άρα παρακολουθούσαμε εμείς εθνικοί βουλευτές πάρα πολύ κοντά, από πολύ κοντά, τη σχετική αυτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Και η Δική Επιτροπή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και πολλές φορές διοργανώνουν και κοινέ συνεδριάσεις των επιτροπών μας. Η πρόεδρος τώρα ζήτησε το λόγο σύντομα για μια παρέμβαση. Το είπε και ο Μάρκα Έντζελε, κύριε Μακάβα, στο τέλος. Πράγματι, στη συνέντευξη υπήρχαν κάποια επίμαχα σημεία και στις δικές μας συζητήσεις εδώ. Δεν είναι η συνένεση όμως ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπή ούτε δική μας του Κοινοβουλίου. Είναι ένα έγγραφο το οποίο διαπραγματεύτηκαν 28 κυβερνήσεις και οι ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάποιε από τις κυβερνήσεις εξέφρασαν θέσεις που δεν μας άρεσαν. Ειλικρινώ το λέω αυτό. Έπρεπε όμως να υπάρξει ένα συμβιβασμό. Επίσης οι υπουργοί έρχονται στις συναντήσεις, προβάλλουν τις εθνικές θέσεις και κανονικά νομίζω ότι μετά πρέπει να ακολουθούν συζητήσεις και στα Εθνικά Κοινοβούλια σε σχέση με την τοποθέτηση του εκάστοτε υπουργού σα και δεν μένει εδώ το θέμα. Σίγουρα και οι εθνικοί βουλευτές έχουν το λόγο Κυρία Έλλης τώρα το λόγο. Thanks, Chair. Uh, colleagues. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντικό που έχουμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψει με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα έχουμε μια κρίσιμη σημασία ευθύνη. Η Ευρώπη οφείλει να δώσει το καλό παράδειγμα σε αυτή την προσπάθεια υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να ηγηθεί. Αν δεν τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι αυτοί οι στόχοι απλώ θα μείνουν στα χαρτιά. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι σήμερα η πολιτική κατάσταση παγκοσμίω είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που είχαμε το 2015 όταν ε, στη Νέα Υόρκη, στα, στον ΟΗΕ, εγκρίθηκαν αυτοί οι στόχοι. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στο τι μπορούμε εμείς να κάνουμε σε αυτή την προσπάθεια. Σύμφωνα με την Concord, η οποία εξέταξε ε, τη, διαδικασία που είχε ακολουθηθεί στα διάφορα κράτη-μέλη. Δέκα χώρες έχουν έναν διαρθρωμένο διάλογο ε, στον οποίο συμμετείχαν και τα Υπουργεία τους για την ε, εφαρμογή αυτών των στόχων. Στο θεσμικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ξεκάθαρο εάν λειτουργεί αυτή η συνεργασία και πρέπει να βρούμε τρόπους να, μην υπάρχει, να, να, σταματήσει ο μεταξύ των Υπουργείων αυτή ε, συζήτηση κατά μόνας. Και όπως πολύ σωστά ε, υπόθηκε, ε, το ζήτημα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, είναι το μέλλον των παιδιών μας. Επομένως, θα πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχουν πολλέ άλλες επιτροπές, όχι μόνο η Επιτροπή Ανάπτυξης, ώστε να υπάρχουν επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να μην γνωρίζουν τη σημασία που θα έχει η δική του συνεισφορά στην παρακολούθηση και την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν πόλεις ε, και περιοχέ, όπω η Κοπενχάγη, οι οποίε έχουν αναπτύξει δικό του τοπικό σχέδιο χρειάζεται να φροντίσουμε την καταπολέμηση των αποκλεισμών με νομοθετικά μέτρα, με προϋπολογισμούς, αλλά και φροντίζοντας να λογοδοτεί η εκάστοτε κυβέρνηση εθνικά και παγκοσμίω. Από τις χώρες όμως οι οποίες, τις οποίες εξέτασε αυτή η μελέτη, μόνο τρία εθνικά κοινοβούλια έχουν κάποιο ε, κάποια ξεχωριστή ομάδα εργασίας, η Φιλανδία, η Γερμανία και άλλη μια χώρα. Θα ήθελα να ζητήσω από τα, τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να πιέσουν έτσι ώστε να δημιουργηθούν τέτοιες επιτροπές. Και κάτι τελευταίο. Από την αρχή της συζήτηση αυτής ζητείται να υπάρξει μια συνολική στρατηγική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να έχει ένα χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένους στόχους. Δεν αρκεί να έχουμε 29 διαφορετικά ε, σχέδια εφαρμογής. Πρέπει όλα αυτά να συντονιστούν μεταξύ τους. Και ε, μια τελευταία παρατήρηση για αυτό που είπε η κυρία Χουίτφελτ από την Νορβηγία η φοροαποφυγή από χώρες αναπτυγμένες είναι ένα τραγικό φαινόμενο. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι, έναντι το οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε. Πρέπει να βρούμε τρόπους καταπολέμησης της φοροαποφυγής η οποία εκτιμάται ότι αποστερεί ε, ε, ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από εθνικούς πόρους που δεν έχουμε στη διάθεσή μας για να τους χρησιμοποιήσουμε για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε κυρία Σλάιν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Στέλλα Μπιάνκη από την Ιταλία. Uh, Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση. είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι αυτό, αυτοί οι στόχοι έχουν τεθεί για όλες τις χώρες, όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες, αλλά και για τις λεγόμενες αναπτυγμένες, που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να εφαρμόσουμε αυτή, το, αυτό το θεματολόγιο, αυτή την ατζέντα η οποία καλύπτει και επηρεάζει όλες τις πτυχές της ζωής κάθε πολίτη, την καθημερινότητά του. Χρειάζεται λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση, μια δομημένη προσέγγιση και μια βηματική προσέγγιση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ιταλία. Ιταλία. Να θέσουμε στόχους σταδιακά, τους οποίους να παρακολουθούμε καθώς εξελίσσονται, καθώς εφαρμόζονται. Επίσης αναφέρθηκε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλληλεπιδράσεις, σχέσεις του κάθε στόχου με τους υπόλοιπους. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, στην εφαρμογή του, του πλάνου. Και τέλος, πιστεύω ότι έχουμε ηθικό χρέος να ξεκινήσουμε από τον στόχο 1, την καταπολέμηση της ε, φτώχειας και την, ε, τον στόχο 2, την καταπολέμηση της πείνας. Έχουμε μείνει πίσω, πίσω εδώ. Και θα πρέπει να το υιοθετήσουμε ως στόχο αυτό και στο εθνικό επίπεδο. Να μην καταπολεμήσουμε την, την, την ε, φτώχεια και την πείνα. Ένας άλλος ε, στόχος, ένα άλλο θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η κλιματική αλλαγή την οποία θα πρέπει να την λαμβάνουμε υπόψη μα σε κάθε πολιτική απόφαση που λαμβάνουμε καθημερινά ε, όσον αφορά τις πολιτικές μας για την ενέργεια, όσον αφορά τις πολιτικές μας για τα συστήματα παραγωγής. Ε, είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να ζούμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη και ειρηνικά. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα να είναι στο, στη, στη, στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χρέος ε, να πετύχουμε το στόχο που ε, αναλάβαμε, τη δέσμευση που αναλάβαμε με τη Συμφωνία των Παρισίων, να φτάσουμε σε μηδενικέ εκπομπέ μέχρι το 2050. Ε, αυτή η συμφωνία δεν είναι απλώ ένα χαρτί. Είναι κάτι που είναι απολύτω απαραίτητο για να επιβιώσουν μικρέ νησιωτικέ χώρε και όλοι μα και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Η ισότητα των δύο φύλων, η ενδυνάμωση των γυναικών είναι πολύ σημαντική και στι αναπτυγμένε χώρε και στι χώρε μα στην Ευρώπη και στι αναπτυσσόμενες χώρε. Ε, αυτό σημαίνει κοινωνική πρόνοια, ε, βοήθεια στι οικογένειε, ε, στα παιδιά. Κλείνω. Ευχαριστώντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων θα πρέπει να αυξάνεται, να συμμετέχουν όλο και περισσότερο μετά την παρουσίαση των Εθνικών Στρατηγικών και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστούμε Στέλλα, λέει η Πρόεδρος. Ο συνεισηγητής, ο κύριος Νόιζερ, ζήτησε το λόγο. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Πολύ σύντομα. Κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό που είπε η Στάμψη από την Ισπανία. Πραγματικά υπήρχε και το παραλαμβάνω σαφής πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Το αποτέλεσμα όμως το οποίο πετύχαμε ήταν ε, σε συνάρτηση και με το τι πέτυχαν τα κράτη-μέλη. Γιατί τα κράτη-μέλη ε, πράγματι είχαν τοποθετηθεί διαφορετικά ξεκάθαρα σε σχέση παραδείγματος χάρη με το στόχο του 0,7%. Ήταν ξεκάθαρο και το λέω για την Ουγγαρία για παράδειγμα. Είπαν ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να μας λένε οι Βρυξέλλες ότι θέλουμε 0,7. Θέλουμε να το αποφασίζουμε εμείς στις ε, χώρες μας. Θέλουμε να το αποφασίζουμε συγκεκριμένα στη Βουδαπέστη εμείς. Και άρα τα πράγματα ήταν δύσκολα εκεί. Το δεύτερο, συνάδελφος από την Νορβηγία που ρώτησε για τη φυγή κεφαλαίων και τη φορολόγηση. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αυτό πρέπει να δώσουμε αποτελέσματα εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο εντός στην Ευρωπαϊκή, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε ό,τι αφορά τις ελίτ, τις αφρικανικές ελίτ. Θα πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Η φοροαποφυγή και η μεταφορά πιστώσεων χρημάτων σε φορολογικούς παραδόσους, παραδείσους είναι κάτι που δεν πρέπει να είναι δυνατόν. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αναφερθεί και να συζητηθεί και στην Αφρική. Δεν θα πρέπει να το αποφεύγουμε, αλλά θα πρέπει να στείλουμε ένα χειρομήνυμα. Τώρα, από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, στον συνάδελφο που μίλησε. Πράγματι υπάρχει αυτή η ε, συνεργασία ε, και στο Αμπιτζάν έχουμε την επόμενη εβδομάδα τη διάσκεψη. Αλλά έχουμε και την κοινοβουλευτική ε, συνέλευση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 28 χώρες ΑΚΕ και 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι αυτή, αυτό το νούμερο έχει και την πλειοψηφία και στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Άρα υπάρχει συνεργασία και μπορεί να έχει αποτελέσματα. Για το συνάδελφο του το Λουξεμβούργο Πράγματι υπάρχουν στη Γερμανία αυτές ε, οι θετικές εξελίξεις για την κλιματική αλλαγή, μετανάστευση ε, που δεν ήταν θέμα ε, που οι συνένεση κατά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ επίσης και για αυτό που είπατε, για την πολύ καλή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό του Λουξεμβούργου, ότι συμμετέχει στο κοινοβουλευτικό έργο κοινωνία των πολιτών και πράγματι θέλουμε μια διπλή στρατηγική να εφαρμόζεται. Δηλαδή θέλουμε και εμείς εδώ την στήριξη από τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί εσείς είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή του 07, αλλά και εσείς από τη δική σας πλευρά ε, θα πρέπει να αναλάβετε τη σχετική δέσμευση και να μας βοηθήσετε και εμάς εδώ ε, σε συνεργασία και σχέση με τα άλλα για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλιούμα Μαμά του Κόντε από το Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, επί τη ευκαιρία που προσφέρετε τη δυνατότητα να λάβει το λόγο το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο να σας ευχαριστήσω και εν ώψη και της ε, Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αφρικανικής Ένωσης ε, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη. Όπως ανέφεραν οι προλαλήσαντες, η νέα κοινή αντίληψη βοηθά να έχουμε ένα βιώσιμο κόσμο στον οποίο θα υπάρχει μεγαλύτερη ευημερία. Και μάλιστα το 2015 όταν η διεθνής κοινότητα ενέκρινε το πρόγραμμα για το θεματολόγιο του 2030 και τις ε, βιώσιμους στόχους για την ανάπτυξη, ε, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η εξάλληψη της φτώχειας ε, και η καταπολέμηση της παγκοσμίω έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη της αυτή τη θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις. Για την Αφρική αυτό σημαίνει εκρίζωση της φτώχειας, αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, εκρίζωση της παράνομης μετανάστευσης, ε, ε, προστασία του περιβάλλοντος, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ούτω καθεξής. Για να μπορέσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτούς τους φιλόδοξους στόχους, αυτή η κοινή αντίληψη θα πρέπει να βασίζεται και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και στο εξή, στη νεολαία, στην ισότητα ανδρών και γυναικών, στην κινητικότητα και τη μετανάστευση, βιώσιμη ενέργεια και κλιματική αλλαγή, επενδύσεις και εμπόριο, καλή διακυβέρνηση και δημοκρατία και κινητοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων. Όλα αυτά ε, σημαίνουν ότι το Παναφρικό Κοινοβούλιο δεσμεύεται για τα όσα τον αφορούν για να μπορέσει να υλοποιήσει και να εφαρμόσει τις μελλοντικέ πολιτικές οι οποίες ε, θα ε, εκπονηθούν για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων και θα λάβει υπόψη της και του παράγοντε αυτού στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφαρμογή του Σχεδίου οικονομική ε, και κοινωνική ανάπτυξη, το 5 ε, το οποίο εκπώνησαν οι Αφρικανικέ χώρε και υπάρχουν συγκεκριμένε δεσμεύσει στον προπολογισμό για την υλοποίηση του προγράμματο, ήδη κατά την άποψή μου αποτελούν μια πρώτη δοκιμή για την συνεργασία μεταξύ ε, Αφρικής ε, ε, Διεθνών Οργανώσεων και του κόσμου των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κοντέ. Και τώρα η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι γίνεται αυτή η κοινή συνεδρίαση, διότι από κοινού μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η νέα κοινή αντίληψη θα είναι ε, κάτι παραπάνω και όχι απλώς ε, κενό γράμμα και ωραία λόγια. Η δική σα δουλειά φυσικά από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι να είναι υπόλογα τα κοινοβούλια σα και να φροντίσετε η κοινωνία των πολιτών να είναι ενήμερη. Ορισμένε φορέ πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών είναι καλύτερα ενημερωμένη από οποιονδήποτε βουλευτή και τους υποφαινόμενους φυσικά περιλαμβάνουν και αυτό είναι θετικό μάλλον. Και επίσης ε, ε, θεωρούμε ότι πρέπει να είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπόλογη και αυτό είναι δική σας δουλειά και θα ήθελα να σταθώ σε κάποια πράγματα χρηματοδότησης. Τώρα, όπως γνωρίζουμε, προετοιμαζόμαστε όλοι για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, που θα ξεκινήσει από το 2021. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να κατανοήσουμε επί ποιες βάσεις ε, προγραμματίζει τα επόμενα βήματά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως δεν θα υπάρξει ε, καμία άλλη τέτοια δυνατότητα για εξειδικευμένα αναπτυξιακά μέσα. Και μπορεί να ακούγεται καλό αυτό, ε, αν υπάρχει το θεματολόγιο για το 2030 και υπάρχει συνεκτική πολιτική για την ανάπτυξη και υπάρχει συνεχώς αυτό το αίτημα. Αλλά ε, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και το γεγονός ότι ορισμένες φορές αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και η αναπτυξιακή στόχοι ε, υπόκεινται σε άλλους στόχους. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην ασφάλεια και στη μετανάστευση και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι εμείς ως στόχο έχουμε να υπερασπιστούμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα να ζητήσω ε, την εξή διευκρίνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι δυνατότητες υπάρχουν ε, για τα διάφορα μέσα και τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη στο νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίση, ε, θα ήθελα να πω ότι ακούσαμε πάρα πολύ καλές ε, παρεμβάσεις από τις χώρες, ε, από τα κοινοβούλια που αποτελούν και υπόδειγμα για την χρηματοδότηση της ανάπτυξη. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απολύτως με το όσα είπε η Ιταλίδα συνάδελφο, που αναφέρθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης για το κλίμα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπερβούμε τους στόχους που έχουμε θέσει, ιδίως τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν ουσιαστικά τη συμβολή τους ε, στη χρηματοδότηση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες και επομένως επαφείται όλο και περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους δωρητέ από τις ευρωπαϊκές χώρες να αντισταθμίσουν αυτό το έλλειμμα, όπως πρέπει να αντισταθμίσουμε και αυτό το έλλειμμα ε, δημοκρατίας του κυρίου Τραμπ που θέτει ε, φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας και γυναίκες σε ε, πολύ μεγάλο κίνδυνο όσον αφορά τα αναπαραγωγικά τους δικαιώματα και τη σεξουαλική τους υγεία. Τέλος, να δώσουμε το λίγο στον Ρόιτ Ράσελ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχει καταρτιστεί μια στρατηγική συντονισμένη για την επίδευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξη. Χάρηκα και που άκουσα προηγουμένως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεισφέρει στην έκθεση και στην παρακολούθηση που θα γίνει με τη συνάντηση της Βιέννης το 2019. Η Επιτροπή Αναπτυξιακής Συνεργασίας στην Βουλή των Κοινοτήτων έχει ε, ζητήσει να συμμετέχει και να παρακολουθεί το θέμα ε, από τη Βρετανική κυβέρνηση. Έχουμε σχεδόν καλύψει το μισό της διαδρομής και όταν πλέον η Ευρωπαϊκή ε, ε, Ένωση εκδώσει τη δικιά της έκθεση θα έχει κλείσει ο πρώτος κύκλος και θα ξεκινάει ο δεύτερος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πολύ ξεκάθαρα και πολύ συγκεκριμένα θα πρέπει να δούμε ποιες περιοχές πολιτικής σε ποιε περιοχέ πολιτική θα δώσουμε προτεραιότητα. Αυτή είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά δεν πρέπει να την καθυστερήσουμε. Γιατί χρειάζεται, για να είναι απολύτω απαραίτητη για να κατανεμηθούν σωστά οι πόροι. Όπω είπαν και πολλοί συνάδελφοί μου εδώ. Είναι λυπηρό ότι αυτή η φοβερή ανανέωση των στατιστικών στοιχείων την οποία μας είχαν ε, υποσχεθεί με την νέα στρατηγική δεν ευοδόθηκε τελικά, δεν έγινε. Στατιστικά στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία θα μας έδιναν τη δυνατότητα να, να, να δούμε ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τις διακρίσεις με βάση την εθνότητα ε, όταν έχουμε μια ολόκληρη κοινωνική ομάδα ή μια εθνοτική ομάδα η μια αθλητικη ομαδα υφίσταται διακρίσεις στο Βρετανικό Κοινοβούλιο ε, έχουμε σκοπό να ξεκινήσουμε μια επιτροπή για να εξετάσει το ζήτημα αυτό. Επίσης θα συμφωνήσω με την αναφορά στην ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή και την μεταφορά κεφαλαίων. Και δική μου την πλευρά και από το δικό μου πολιτικό κόμμα αυτό που θα πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, η Βρετανία θα πρέπει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια, αντί να περιμένουμε οι αναπτύσσόμενε χώρε να ε, ηγηθούν τις προσπάθειες καταπολέμησης της φοροαποφυγής. Αν δει κάνει τα έγγραφα του Παναμά, οι χώρε που βρίσκονται, που, αναφέρονται, οι εταιρείε που, πρωτοστατούν στην φοροαποφυγή είναι ευρωπαϊκέ και Αμερικανικέ. εάν δεν υπήρχαν τέτοιου τύπου πρακτικές και ε, ε, δινόταν η δυνατότητα στι αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τη δική τους φορολογική βάση, θα φτάναμε σε ένα σημείο που δεν θα χρειαζόταν καν η άμεση αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα κλείσουμε τα παραθυράκια, ε, είτε αυτά είναι στο εσωτερικό της Ένωσης, όπως το City του Λονδίνου, του Λουξεμβούργου, είτε βρίσκονται εκτός όπως η offshore και άλλες φορολογική παράδειση. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ ξεκάθαροι και να αναλάβουμε σοβαρή δράση. Δεν αρκεί απλώς να το αναφέρουμε στα, στα λόγια. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της φοροαποφυγής ε, αν ε, υπερισχύει πάντα η προσπάθεια να βρούμε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του 0,7 του ΑΕΠ, όμως γίνεται όλο και δυσκολότερο ε, σε εθνικό επίπεδο να το υπερασπιστούμε αυτό και να το πετύχουμε όταν υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες δεν αναλαμβάνουν και δεν πετυχαίνουν αυτή τη δέσμευση του 0,7%. Στο εσωτερικό της χώρας μου οι πολίτες λένε γιατί εμείς να πρέπει να το κάνουμε όταν οι άλλοι δεν το, δεν το προσπαθούν. Ε, ελπίζω να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να δώσω για ένα λεπτό μονάχα στον εκπρόσωπο τη Επιτροπή το λόγο, τον κύριο Φροντίνη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να απαντήσω σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν στη συνεδρία σε αυτή σε ένα λεπτό. Θα σταθώ λοιπόν σε δύο ζητήματα που συζητήθηκαν πολύ. Πιστεύω ότι είναι άδικο να λέει κανείς ότι η κοινή αντίληψη, η νέα, ε, δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία στην καταπολέμηση της φτώχειας. Αντιθέτως. Όμως, αντιληφθήκαμε με την προηγούμενη ατζέντα ότι είναι αδύνατο να καταπολεμήσει κανείς την φτώχεια αν δεν ε, αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή, τις ανισότητες, την σταθερότητα οι χώρες εκείνες στις οποίες σημειώθηκε η μικρότερη πρόοδος όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας ήταν εκείνες οι χώρες οι οποίες βρίσκονταν σε, κρίση. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αντιστοίχως, η μετανάστευση είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ε, είναι μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτό φαίνεται στην ε, κοινή αντίληψη. Βέβαια, όπως σωστά ελέγχθη, όταν ε, προσπαθεί κανείς να βρει ε, μια κοινή αντίληψη, ένα συμβασμό στον οποίο να συμφωνούν 28 κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χρειάζεται να γίνουν αμοιβέ παραχωρήσεις. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να φαίνεται ε, και να συνεχίζεται ε, αυτή η δέσμευση των ευρωπαϊκών κρατών στο 0,7% του ΑΕΠ τους για την ανάπτυξη. Πολύ λίγες χώρες το έχουν πράξει αυτό. Και χρειάζεται ένας μηχανισμός παρακολούθησης. Όπως είπα το 2019 θα πάμε στα Ηνωμένα Έθνη και θα παρουσιάσουμε μια έκθεση στην οποία θα φαίνεται με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαϊκές χώρες εφάρμοσαν ε, το θεματολόγιο αυτό, αυτούς τους στόχους. Και πιο συγκεκριμένα, ποιες χώρες έφτασαν και πέτυχαν το 0,7%. Ε, ίσως να μην έχουμε ένα σύστημα τέλειο ή όσο ανεπτυγμένο θα θέλαμε. Αλλά πάντως υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα παρακολούθησης. Σας ευχαριστούμε κύριε Φροντίνη. Στο συγγνώμη δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε αυτό, ε, στη σημείο σε άλλους σας ευχαριστώ. Τι. Η κυρία Χάουτελα. Ναι, αλλά θέλουμε να ακούσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέσαμε, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το ζήτημα της χρηματοδότησης, για παράδειγμα. Η πρόεδρο, αυτό σημαίνει όμω ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το δεύτερο γύρο συζήτηση και δεν είναι δίκαιο αυτό. Ζητώ συγγνώμη, ζήτησαν πάρα πολύ το λόγο και ξεπέρασαν και το χρόνο ομιλία του. Είμαι από την ομάδα των φιλελευθέρων ο συντονιστή. και ξέρετε ότι πολλές φορές έχουμε αλληλεπικαλυπτόμενε συνεδράσεις. Άργησα να έρθω και ήθελα κι εγώ να εγγραφώ στον κατάλογο των ομιλητών. Δεν μπορούμε να είμαστε πανταχού παρόντες όμως δυστυχώς γιατί υπάρχουν διάφορες συνεδριάσεις που γίνονται ταυτόχρονα. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μας ε, με τη, τα Εθνικά Κοινοβούλια έχω να πω κάποια πράγματα και ίσως και άλλοι συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να συντομεύσουμε το δεύτερο τμήμα, το δεύτερο πάνελ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όσοι θέλουμε. So, Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Δεν έχουμε όμως χρόνο ούτε για ερωτήσεις ούτε για άλλες παρεμβάσεις. Όσοι πάντως έλαβαν το λόγο νομίζω ότι ε, κατέστησαν σαφές πόσο σημαντική είναι η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την επιτυχία των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες ιδίως και ελπίζω να αποτελέσει αυτή η συνένεση το σημείο αναφοράς για πολιτικές και νομοθετικές αποφάσεις σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος, το πρώτο τμήμα της μερίδας και περνάμε στο δεύτερο πάνελ. Η Λόλα θα προεδρεύσει. Αυτά από πλευρά μου. Σας ευχαριστώ. Hi. We need to start. Can you please take your... Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε. Venga, pues empieza I will speak in Spanish. Θα μιλήσω ισπανικά. Bueno, muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Λόλα Σάντσεφ Καλτεντέ, είμαι μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι από την Ισπανία, εκπροσωπώ το Ποδέμος, το οποίο συμμετέχει στην ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, την ΚΟΕ. Στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης θα συζητήσουμε τις προοπτικές για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για την ε, ε, συγκεκριμένη στόχευση αυτής της ε, συνεδρίασης. Ο στόχος δεν είναι να προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε τις δεσμεύσεις και την πρόοδο στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Αντιθέτως, θέλουμε να δούμε τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη μέσω της εξωτερικής πολιτικής και της βοήθειας για την ανάπτυξη για να προωθήσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η έγκριση αυτών των στόχων το Σεπτέμβριο του 2015 αποτέλεσε αλλαγή στην προοπτική της πολιτικής ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Στο παρελθόν, οι στόχοι της χιλιετίες ε, προσπαθούσαν να κρυζώσουν την παγκόσμια φτώχεια και ήταν υπέρ ε, μια σχέσης ε, δωρητή δικαιούχο. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης προωθούν ένα παγκόσμιο θεματολόγιο, στην οποίο οι αναπτύσσόμενε χώρες και οι χώρες υποανάπτυξη ανάπτυξη ε, είναι υπεύθυνε για την εκτέλεση και των στόχων, όπως και οι υπόλοιποι ε, που συμμετέχουν στην ανάπτυξη. Η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης, λοιπόν, ε, μας θέτει όλους υπεύθυνου και πρέπει να αλλάξουν οι ισορροπίες σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, με στήριξη από ολοκληρωμένε πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανάπτυξη μέσω σωστών διαδικασιών καλής διακυβέρνησης, με εστίαση στην συμμετοχή πολιτών. Γι' αυτό ακριβώ και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επισημάνουμε την ε, ε, ε, αρχή της δημοκρατικής εξοικείωσης. Θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια και τα πολιτικά κόμματα, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, η κοινωνία των πολιτών και όλοι όσοι συμμετέχουν να ε, συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δύο χρόνια μετά την έγκριση των SDG πρέπει να γίνει ε, μια, ένας απολογισμός του που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούμε κατά πόσον οι στρατηγικές πολιτικές και οι δομές ε, διακυβέρνησης υπάρχουν και αν έχουν καθοριστεί κατάλληλοι μηχανισμοί ε, για ε, την ανάληψη ευθυνών. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε καλέσει τον κύριο Γκουίντο ε, Σμιτ Τρόου, εκτελεστικό διευθυντή του δικτύου βιώσιμων αναπτυξιακών λύσεων που θα παρουσιάσει τον δίκτυ και τον κατάλογο των μέσων του 2017 που εκπονέθηκαν από το δίκτυο. Έχετε το λόγο κύριε Σμιτ Τράουμπ για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα για να μοιραστώ κάποιε σκέψει για το τι γίνεται με την εφαρμογή των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μαζί με του συναδέλφου μα ε, ε, προσπαθούμε να δούμε, στον Bertelsmann Stiftung, προσπαθούμε να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε καλύτερα στοιχεία, περισσότερα στοιχεία, ώστε να μπορούν να κάνουν και καλύτερο απολογισμό τη κατάσταση στα κοινοβούλια. Γνωρίζουμε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι κρίσιμη σημασία για τους δημοσίου διαλόγους στι αναπτυσσόμενε χώρε, όπως ε, τόνισαν οι πρόεδροι, αλλά και στις ανεπτυγμένε χώρες. Και αυτό που χρειαζόμαστε σίγουρα είναι μια πιο ισχυρή συζήτηση για τα θέματα αυτά, διότι οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν είναι ε, βαθιές ε, και δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να μπούμε στη σωστή οδό για να τι επιτύχουμε. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε καταρχώς τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την δράση πολιτικής. Όχι απλώς ένα εργαλείο λοιπόν που συζητούν οι ειδικοί στις αρμόδιες επιτροπές, αλλά να το εξετάσουμε ευρύτερα στους στόχους πολιτικής. Με ενθαρρύνει ε, πολύ ε, ο τρόπος με τον οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί οι στόχοι, πολύ περισσότερο από τους στόχους της χιλιετίας στους οποίους συμμετείχα, αλλά κυρίως πρέπει να αυξήσουμε την ενημέρωση. Πρέπει να γίνουν ε, εθνικές συζητήσεις για τις προτεραιότητες τη θέση στόχων και τη διαμόρφωση των στρατηγικών εφαρμογής ε, των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, ε, θα πρέπει να έχουμε επίσημες δείκτες ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Προχωρά αυτή η δουλειά, αλλά είναι περίπλοκη και από τεχνική σκοπιάς και ε, ε, δυσχεραίνεται και λόγω της διαθεσιμότητας των στοιχείων. Τι κάναμε εδώ. Εδώ έχουμε ένα απόσπασμα και θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία τα οποία λάβαμε υπόψη. Χρησιμοποίησαμε τα ε, διαθέσιμα στοιχεία για να δούμε πού βρίσκονται οι χώρες γενικά. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα απόσπασμα της βαθμολόγησης των στόχων βιώσιμης απο... Ανάπτυξης και βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες στείλουν να βρίσκονται στην κορυφή των δικτών. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν πολύ σημαντική επιτυχία για την Ευρώπη, διότι ουσιαστικά είναι σαν ο κόσμος να προσυπογράφει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο σε όλες τις χώρες που έχουν οικονομία κοινωνικής αγοράς με περιβαλλοντική ε, βιωσιμότητα. Υπάρχουν φυσικά διαφορές ε, ε, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ε, το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεν είναι το μοντέλο των ΗΠΑ και σίγουρα όχι της Κίνας. Ε, η Ευρώπη τα πηγαίνει σε γενικές γραμμές καλά, σε συνολικό βαθμο, σε συνολική βαθμολογία έχουμε περίπου 83 δείκτες, το 100 είναι το βέλτιστο και το 0 φυσικά σημαίνει ότι είστε στο ναδύρ τη κατανομής ε, όσον αφορά τα απόλυτα πρότυπα. Τι θέλουμε να επιτύχουμε λοιπόν για τη μείωση των στόχων, ε, για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου κλπ. Εδώ υπάρχει και το εξή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε βρίσκονται στην 42η θέση, που αποτέλεσε και έκπληξη για την άλλη πλευρά του αποκλατικού, αλλά οφείλεται κυρίω στο γεγονό ότι επειδή υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό ε, εισοδήματο, υπάρχουν πολύ ψηλά ποσοστά παιδική θνησιμότητα, ε, πολύ ψηλά επίπεδα βία, ε, υψηλέ ανισότητε και από περιβαλλοντικέ σκοπιέ, βέβαια, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία. Πολλά μπορούν να γίνουν και θα μπορέσω να ε, εξηγήσω και κάποια πράγματα. Ε, επικεντρωθήκαμε σε αναπτυσσόμενες χώρες, ε, αλλά θα δείξω και κάποια στοιχεία για ευρωπαϊκέ χώρε. Εδώ έχουμε το παράδειγμα τη Ινδονησίας. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι λεπτομέρειε, αλλά η Ινδονησία βρίσκεται στο 100 από τι 157 χώρε που εξετάσαμε. Στη μέση έχουμε άλλα ε, αναπτυξιακά μέτρα. Η Ινδονησία πηγαίνει πολύ καλύτερα στην παγκοσμία ανταγωνιστικότητα ε, είναι σημείο λοιπόν στο οποίο έχουν θέσει ως προτεραιότητα και πηγαίνει πολύ καλύτερα στο ΑΕΠ κατά κεφαλήν, αλλά ε, συνολικά οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ε, έχουν μια σειρά από προκλήσεις που δεν έχουν αποσχολήσει τόσο πολύ αποτελεσματικά τη χώρα. Ε, το ίδιο βέβαια μπορεί να ισχύσει και για ευρωπαϊκές χώρες. Ε, στο κάτω δεξιά σημεία βλέπουμε αναστόχο ποιο είναι το μέσο ε, επίτευμα. Αν δείτε την κάτω στήλη λοιπόν εδώ έχουμε τους στόχους στους οποίους έχουμε βασικές προτεραιότητες πολιτικές και υπάρχουν μεγάλα κενά εφαρμογής και υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέτρα στα οποία η χώρα ε, έχει κακή βαθμολογία. Για παράδειγμα ε, υπάρχει ε, κακή διατροφή και υποσυτισμός αλλά υπάρχει και αυξημένο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ινδονησία. Εδώ έχουμε ε, την απόδοση 20 χωρών, ε, έχουμε τις χώρες του G20 εδώ, δεν φαίνονται βέβαια πάρα πολύ καλά, έχουμε επάνω τις χώρες εκτός ΟΣΑ και από κάτω έχουμε τις χώρες, του ΟΣΑ που, είναι, ε, τις χώρες συγγνώμη, που είναι μέλη του ΟΣΑ, έχουμε εδώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το βασικό είναι ότι υπάρχουν πολλά κόκκινα που σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα τα οποία δεν εμφανίζονται παρκώς στις εσωτερικές συζητήσεις. Πολλά στοιχεία θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σα και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να τα βρείτε χρήσιμα για την αξιολόγηση τη ε, συνεισφορά τη χώρα σα, για να δείτε αν υπάρχουν τομείς στους οποίου θα μπορούσατε να τα πάτε καλύτερα. Ο στόχο 17 που είναι ο δεξιά, οι διεθνεί εταιρικέ σχέσει, βλέπετε ότι έχουμε πολλά κόκκινα και μεταξύ των κρατών μελών. Ε, θέματα που αφορούν φορολογικούς παραβα... Ε, παραδείσους, ε, τραπεζικό απόρριτο κλπ. Και εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτή της δουλειάς. Αυτό το διάγραμμα ε, κάτω, οριζόντια, έχει το ΑΕΠ ε, ε κατά κεφαλή, ε, επομένως έχουμε τις πλουσιότερες χώρες και στον κάθε το άξονα έχουμε τις ε, παράπλευρες επιδράσεις. Ε, τι μπορούμε να έχουμε, για παράδειγμα, σε περιβαλλοντική πολιτική, ε, σε οικονομικές πολιτικές, σε ασφάλεια για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν πολύ κακή βαθμολογία. Πάνω πάνω έχουμε την Ελβετία, δεν είναι χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε την Κύπρο, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο, που έχουν άσχημες επιδέσεις και πολλές διακυμάνσεις. Η Δανία και η Ισλανδία βρίσκονται πολύ κάτω ε, για αντίστοιχο επίπεδο εισοδήματος. Υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα τα οποία δεν ε, αντιμετωπίζονται καταλήλως και υπάρχουν και ε, σημαντικές συνέπειες και αυτά είναι σημαντικά. Το ίδιο μπορούμε να το δούμε και σε ε, κατακαιρματισμό σε εθνικό επίπεδο. Είδαμε τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, τι γίνεται σε επίπεδο πολιτείας και πόσο ισχυρή είναι η στόχη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι κόκκινες ε, περιοχές είναι οι περιοχές στις οποίες είχαμε τις μεγάλες αλλαγές στις τελευταίες εκλογές, μεγάλες αναταραχές επίσης, ε, υπάρχουν οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο πλαίσιο για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Κάποια επόμενα βήματα τώρα, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είναι χρήσιμο και αυτό. Δημοσιεύουμε μια επόμενη έκδοση το καλοκαίρι του έτους. Ε, έχουμε στοιχεία για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στην έκθεση. Θα εξετάσουμε και τις τάσεις για πρώτη φορά για να δούμε αν είστε στο σωστό ή στο λάθος δρόμο. Έχουμε και κάποια στοιχεία τα οποία λάβαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Εξετάζει εξετα... Ε, τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες νέες μορφές δεδομένων. Εξετάζουμε τι κάνει κάθε χώρα για να εφαρμόσει και να βελτιώσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, βλέπουμε τι γίνεται ε, σε κάθε χώρα και επίσης θα δούμε και περιφερειακούς δείκτες. Θα ξεκινήσει ένας δείκτης με χώρες της Αφρικής, ε, εξετάζουμε αφρικανικές οικονομίες τις χώρες ΑΣΕΑΝ, η Κίνα για παράδειγμα ε, θα μπορούσε να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη και βλέπουμε και σε ευρωπαϊκό ίσως πλαίσιο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, τι κάνει η Eurostat. Προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα για τους δείκτες για τις πόλεις και ε, ένα δείκτη για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Υπάρχουν λοιπόν πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, κάποια χρησιμοποιούνται, αλλά πολλά από αυτά τα οποία ε, βρίσκουμε και διαπιστώνουμε δεν είναι γνωστά στις κυβερνήσεις και θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σμιτράουπ. Τώρα, η κυρία Κέιτ Πέντους Ρωσιμάνους, αντιπρόεδρος ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ε, του Εσθονικού Κοινοβουλίου. Η Εσθονία έχει την εκπεριτροπής προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής για το εξάμεινο αυτό. Παρακαλώ, Κέιτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, αξιότιμοι βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να σα ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η Επιτροπή σας ε, για να παραμείνει στο επίκεντρο η πρακτική υλοποίηση των πολιτικών δεσμεύσεων ε, και η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει πραγματικά σε αυτούς που περισσότερο τη χρειάζονται, νομίζω είναι πραγματικά σημαντικός. Ίσως ε, δεν υπάρχουν πολλοί που αμφιβάλλουν ακόμη για το ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης είναι ορθοί, είναι αναγκαίοι, αλλά το πρόβλημα πάντοτε όσοι ήθιστε είναι η εφαρμογή, η υλοποίηση των στόχων. Και μια από τις ανησυχίες που εκφράζονται όλο και πιο συχνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα οξέα εσωτερικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση και να χαθεί η συνολικότερη εικόνα Σίγουρα στα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, πολλοί που συνεχώς θέτουν το ερώτημα γιατί δίνουμε τόση προσοχή πέραν των συνόρων και δεν λύνουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα. Δηλαδή, αν στάζει η οροφή σου, θα κοιτάξεις ε, αν έχει σπασμένο παράθυρο γείτονας θέλει πολύ σθένος ε, βούληση ε, να εξηγήσει κανείς ε, γιατί είναι πραγματικά και προς το δυτικό μας το συμφέρον αλλά και είναι και καθήκον μας να παράσχουμε βιώσιμη αναπτυξιακή βοήθεια και πέραν των συνόρων των εθνικών. Και νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε υπόψη ότι το 85% των Ευρωπαίων πολιτών σήμερα πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους από τις ανεπτυσσόμενες χώρες. Και τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι η βοήθεια προς τις στοχές χώρες θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα πρέπει η Ένωση να τηρήσει τις παρελθούσες δεσμεύσεις της και να τις αναβαθμίσει, μάλιστα. Συζητήσαμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, σε μια εποχή που δεν ήταν πλέον ε, ε, τόσο οξυμένη η χρηματοοικονομική κρίση και δεν είχε οξυνθεί τόσο το, μεταναστευτικό πρόβλημα, που τώρα όμως έχει. Άλλες ήταν οι προκλήσεις που είχαμε αντιμετωπίσουμε τότε. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί οι προκλήσεις και δεν θα λυθούν δυστυχώς ούτε και στο άμεσα προβλέψιμο μέλλον. Υπάρχουν κάποιες μεγάλες τάσεις που θα επηρεάσουν τον κόσμο τα επόμενα 20-30 χρόνια. Και μάλλον θα είναι η κλιματική αλλαγή που αναφέρθηκε, η ταχεία αύξηση του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όλο και πιο πολλά αποτυχημένα κράτη, δημογραφικές αλλαγές κτλ. κτλ. Άρα χρειάζεται καλά συντονισμένη και στοχευμένη υποστήριξη. Και αυτή η ανάγκη θα αυξάνεται και δεν θα περιορίζεται στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα το θεματολόγιο και την επίτευξη αυτών των στόχων, είναι μακροπρόθεσμη στόχη. και σίγουρα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλες τις προεδρίες μέχρι το 2030 και μετά ίσως από το 2030. Άρα καταλαβαίνετε ότι αποτελούν προτεραιότητα και για την Εστονική Προεδρία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Προεδρία μας ε, ήταν υπερήφανη που διοργάνωσε μια παράπλευρη εκδήλωση στο πλαίσιο του ΙΕ για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη ε, στην αλυσίδα αξία ε, στη βιομηχανία τη κλωστοϊφαντουργία. Ένα τεράστιο κλάδο, κλωστοϊφαντουργία, που όμως παράγει τα περισσότερα απορρίμματα και ρήπους. Το 100% των υλικών ε, καταλήγουν ως απόβλητα. Επίσης ε, είναι επιβλαβή σε αυτές δραστηριότητες προς το περιβάλλον. Και ο κύριος Έλιοντ Χάρης είχε πει τότε ότι για να πετύχουμε την εφαρμογή των στόχων ε, βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να περιλάβουμε τους σχετικούς κλάδους. Και όπως είπε, η ένδυση κλωστεφαντουργία είναι ένας από τους τομείς που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους σε παγκοσμίο επίπεδο. Κυκλική οικονομία ε, είναι σημαντική και η προσέγγιση ε, που λαμβάνει υπόψη τον κύκλο ζωής πρέπει να προτιμηθεί. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι Υπάρχει χώρες που εξαρτώνται από αυτόν τον κλάδο, όπως ε, το Μπαγκλαντές, γιατί είναι ο τομέας της ένδυσης των υφασμάτων ε, αυτός ε, που προσφέρει τις περισσότερες εξαγωγές. Άρα και οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις έχουν το ρόλο τους εδώ. Πρέπει να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Άρα, όπου και αν λαμβάνει η χώρα η παραγωγή, θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια βιωσιμότητας. Και εμείς οι αγοραστές πρέπει να επιβρεάζουμε και εμείς τα πράγματα. Ο πρόεδρος, η Τροψικέρα Μακάβαν, έκανε ένα πολύ εμπνευσμένο λόγο. Μίλησε για την εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης στον τομέα της ένδυσης. Μια πρωτοβουλία μετά την, που ήρθε ως απόρρια της καταστροφής στο εργοστάσιο στον Παγκλαντές. Το Φεβρουάριο φέτος ο Σάιν έκρινε κατευθυντήριες γραμμές δεσμευτικές στο σε επιμέλεια και για να κατανοηθεί καλύτερα η αλυσίδα εφοδιασμού. Αλλά όλα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν από κάποιον. Άρα η δική σας αφοσίωση και η δική σας πίεση ήταν κάτι πολύ σημαντικό και το εξηγήσετε και στη Νέα Υόρκη, πολύ ξεκάθαρα. Η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη προσφέρει πολλούς καινοτόμους τρόπους για την προσέγγιση του θεματολογίου του 2030 και σε ό,τι αφορά τη χρήση ψηφιακών λύσεων και τεχνολογιών. Είναι όμως σημαντικό, και υπόθηκε και στην προηγούμενη συνεδρία, ο βασικός, ο πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να παραμείνει η εκρίζωση της φτώχειας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη όχι μόνο να πιέζουν για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά να εφαρμόζουν τους στόχους αυτούς και εσωτερικά, γιατί εφαρμόζονται, ισχύουν για όλες τις χώρες αυτοί οι στόχοι, άρα δεν μπορούμε να πείσουμε άλλους να ε, τους επιδιώξουν αν εμείς δεν το κάνουμε. Έχει ακουστεί πολλές φορές εδώ σήμερα ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να απαντήσει για τα επόμενα 20-30 χρόνια ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα. Πώς θα παραμείνει ανταγωνιστική, πώς θα αυξήσει την ευημερία των πολιτών της. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης σίγουρα δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτό το στόχο αλλά είναι συμπληρωματικοί, συνεπικορούν ε, την επίτευξη αυτού του στόχου. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρκ Τζακομίνη που είναι αναπληρωτής ε, ε, εκτελεστικός διευθυντής για παγκόσμια πολυμερή ζητήματα στην ΕΕΘ. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ λέγοντα ότι η στόχη βιώσιμη ανάπτυξη είναι γενικό στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ταυτίζεται με τι αξίε μα και συνεισφέραμε ε, στην υιοθέτηση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος για το 2030 στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Έχουμε λοιπόν δεσμευτεί και διεθνώς και εσωτερικά να προσπαθήσουμε για να τα πετύχουμε αυτά τα πράγματα μιας και μου ζητήσατε να εστιάσω στο, στη διεθνή διάσταση, δεν θα αναφερθώ στην δουλειά που κάνουμε στο εσωτερικό. Πέρα από το εξή, ε, έχουμε ξεκινήσει τη σύνταξη ενό κειμένου περισυλλογή, ενό κειμένου προβληματισμού που θα δημοσιευθεί στο δεύτερο εξάμεινο για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα το ξεκινήσουμε να το συζητάμε αρχές του 2018 και 28 Νοεμβρίου θα δημοσιοποιηθεί και μια σχετική έκθεση με στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Όπως είπα λοιπόν και προλαλήσαντες, είναι σημαντικό να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ των προσπαθειών που κάνουμε στο εσωτερικό της Ένωσης με τις προσπάθειες που κάνουμε διεθνώς, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ξεκινήσαμε από τα του οίκου μας. Από την πλευρά μας η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι γνωστό ότι πράττει. Έχουμε αναλάβει δράση ως Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή ασφάλεια συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο στο οποίο αναφέρεται η σημασία που έχει η υποστήριξή μας στον ΟΗΕ για τη, για τη διεθνή συνεργασία και οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη έχουν μεγάλη σημασία σε αυτήν την προσπάθεια συνεργασία με τον ΟΗΕ. Έχουμε επίση την κοινή αντίληψη που φτιάχνει ένα νέο πλαίσιο για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη της για την αναπτυξιακή συνεργασία και αυτό το νέο πλαίσιο πολιτικής έχει βασιστεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και δίνει το μήνυμα ότι θα υπάρξει πιο στενή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων μας, των τρίτων χωρών δηλαδή, προκειμένου να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Και ως παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις προσπάθειες που γίνονται για ε, συνεργασία πιο σταθερή, την κατάπτυση χρονοδιαγραμμάτων από κοινού κτλ. την διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία τη βλέπουμε και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο πλαίσιο των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τους, με τις άλλες χώρες, ε, τη σχέση που έχει με την ανθρωπιστική βοήθεια, με τις εμπορικές συμφωνίες, με την πολιτική μας στο, για το κλίμα, για το περιβάλλον. Και τέλος, έχουμε και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Επενδύσεων, το οποίο θα προσπαθήσει να ενισχύσει τις ε, άμεσες ε, επενδύσεις στην Αφρικανική Ήπειρο ε, και το οποίο έχει και αυτό καταρτιστεί επί τη βάση της νέας προσέγγισης μας. Πώς περνούμε τώρα από την στρατηγική στην υλοποίηση. γνωρίζετε στο πλαίσιο της στρατηγικής ότι την, την ευημερία θα πρέπει να την μοιραστούμε ισότιμα όλοι και το αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να επιτευχθούν εξίσου σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης αναγνωρίζετε ότι δεν μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά αν δεν υπάρχει ασφάλεια και ειρήνη έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα, Resilience Initiative, με την οποία προσπαθούμε να έχουμε έναν τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων όπως η φτώχεια, η ε, μετανάστευση, ε, η ε, έλλειψη σταθερότητας Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι κάθε χώρα θα είναι σταθερή, θα είναι ανθεκτική σε κρίσεις, σε προκλήσεις, σε ιδιαίτερες καταστάσεις, έκτακτες καταστάσεις. Για να συμβεί αυτό πρέπει να γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου, να, να υπάρχει προετοιμασία και να υπάρχει μια καταγραφή των διπλωματικών και πολιτικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να κινητοποιούνται κατάλληλα την στιγμή που χρειάζεται. Σας ανέφερα πριν τις προσπάθειες που κάνουμε για την υποκοινού κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων. Έχουμε επίσης ε, ε, μια προσπάθεια για να έχουμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την επιδείνωση της κατάστασης σε κάποιες χώρες όπου υπάρχει τέτοιο κίνδυνος. Είτε πρόκειται για την ανθρωπιστική κατάσταση, είτε για την πολιτική διάσταση κάποιων συγκρούσεων ή κάποιων ευαίσθητων περιοχών. Αυτό το πλαίσιο για την αθεκτικότητα πιστεύω ότι είναι, ε, κάτι που βοηθάει στην πρόοδο την κοινωνική και είναι μια βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη προσέγγιση που είχαμε, όπου εστιαζόταν μόνο στι ευαίσθητε, στι επικίνδυνε, αν θέλετε, χώρε. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζακομίνη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου και όπως ε, είπε και η συνάδελφος προηγουμένως, σας παρακαλώ να είστε πολύ συγκεκριμένοι για να έχουμε αρκετό χρόνο. Θα δώσουμε 2,5 λεπτό λοιπόν, 2,5 λεπτά στον καθένα. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω να συστηθείτε πριν από την ε, παρουσίασή σας ε, το όνομα και τη χώρα καταγωγής σας και αν έχετε κάποια ερώτηση να πείτε σε ποιον την απευθύνετε. Ξεκινούμε με την Ισπανία. Χωσέ Αντώνιο Ρούμπιο, παρακαλώ. Καλημέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο Χωσέ Αντώνιο Ρούμπιο, γερουσιαστής ε, στην Ισπανία. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την διοργάνωση αυτής της διακοινοβουλευτικής ε, συνεδρίασης, για το θεματολόγιο του 2030 που θεωρώ ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να ε, λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική όλων των χωρών για ό,τι κάνουμε τα επόμενα χρόνια διότι από αυτό θα εξαρτηθεί και το μέλλον της ανθρωπότητας. Η γερουσία στην Ισπανία διεξάγει κάποιες δραστηριότητες, κυρίως για ευαισθητοποίηση και για να τεθεί ε, στο προσκήνιο ε, το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, διότι σίγουρα μας απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχει άγνοια μεταξύ αρκετών πολιτικών, αλλά και στην κοινωνία εν γέννη. Ε, και ακριβώς Γι' αυτό το λόγο κάνουμε κάποιες πολύ σημαντικέ προσπάθειες και συστήθηκε και μια ειδική επιτροπή για την εφαρμογή των στόχων βιώσιμη ανάπτυξης στην οποία συμμετέχουν όλες οι δημόσιες διοικήσεις, ε, ε, όλοι οι εκπρόσωποι και η κοινωνία των πολιτών εν γέννη. Και εκεί ε, φάνηκε ότι υπάρχει όντως άγνοια και γι' αυτό ακριβώς ε, και ε, θέλουμε το Φεβρουάριο να γίνει μία συνεδρίαση στην οποία θα συμμετέχουν οι Προεδροί και οι εκπρόσωποι όλων των επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων του ε, Κογκρέσου και της Γερουσίας, καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των ε, Κοινοβουλίων των Αυτόνομων Περιφερειών και των εκπροσώπων της ε, ε τοπικής κοινωνίας από δήμους και επαρχίες, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το θεματολόγιο 2030 και να αξιολογήσουμε και το σχέδιο το οποίο θα υλοποιήσει η Ισπανία τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Μαρία Μανουέλ Ρόλα από την Πορτογαλία. Καλημέρα σας. Αναλύοντας τους δείκτες που παρουσιάζονται σήμερα, είναι απόλυτα σαφές ότι η Ευρώπη ξεχωρίζει, είναι διαφορετική. Αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα και το γεγονός ότι μπορούμε να μεταλαμπαδεύσουμε προς τα έξω και πολλούς αρνητικούς παράγοντες και νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει και ένα επιπλέον θέμα το οποίο θα ήθελα να θέξω που αφορά την Πορτογαλία και την Ισπανία και την ε, Ιβηρική Χερσόνησο και την κλιματική αλλαγή στην Ιβηρική Χερσόνησο. Οι 12, 13 και 14 στόχοι αφορούν το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό θέτει και το ερώτημα πώς μετρούμε την κλιματική αλλαγή, τι παράγοντες πρέπει να ε, υπολογίσουμε. Οι χώρες του δεν έχουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Είναι αρνητικά τα στοιχεία σε αυτούς τους τρεις ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη ε, ανησυχία. Η Πορτογαλία επίσης δεν έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Υπάρχει βεβαίως και το φαινόμενο των ε, δασικών πυρκαγιών που βιώσαμε, ε, υπάρχει μια φρικτή ξηρασία στη Νότια Ευρώπη που δεν φαίνεται ότι θα ε, περάσει σύντομα. Ε, πώς λοιπόν σκοπεύουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα, πώς ε, ε, θα μειώσουμε τη σπατάλη του ύδατος, πώς μπορούν να διοχετεύεται για παράδειγμα τα ύδατα από μια λεκάνη ενός ποταμού σε άλλες χώρες, σε χώρες που δεν ε, ε, έχουν τόσο πολύ ε, μεγάλα αποθέματα υδάτων και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία. Υπάρχει έλλειψη πόρων, υπάρχει έλλειψη πόρων στην Ισπανία που θα επηρεάσει και την Πορτογαλία κατά συνέπεια. Έλλειψη πόρων θα σημαίνει και μεγαλύτερη μετανάστευση και ποιος ξέρει μπορεί να οδηγηθούμε και σε πόλεμο. όλα αυτά τα θέματα λοιπόν πρέπει να τα έχουμε κατά νου όχι μόνο παγκοσμίω αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Θα ήθελα λοιπόν να τα περάσουμε από το τοπικό σε ευρύτερο παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η Σούζαν Κούρς από την Ισπανία, από την Αυστρία, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέγομαι Σουζάνε Κούρτς και είμαι από την Bundesrat, από το Αυστρικό Κοινοβούλιο. Πραγματικά ε, θα πρέπει να αναλάβουμε συνολικά την ευθύνη και η ε, Αυστρία έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη μέσω διαφόρων φορέων. Το ίδιο ισχύει και για την επιτέξη των στόχων ε, του θεματολογίου 2030. Έχουμε αναπτυξιακή συνεργασία, υπάρχουν, ε, υπάρχει συνεργασία με, με όλους τους φορείς για τη μείωση της φτώχειας, τη μεγαλύτερη προστασία της ανθρωπότητας, προστασία του περιβάλλοντος, των πόρων, που είναι πολύ σημαντικοί στόχοι για τη, και αναφέρονται και στο στόχο, στο νόμο τον Αυστριακό για την αναπτυξιακή συνεργασία. Σίγουρα λοιπόν ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Τα θέματα αυτά επάγονται στο Αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε και έναν οργανισμό για την αναπτυξιακή συνεργασία που θεσπίζει προγράμματα και projects σε συνεργασία με δημόσια ιδρύματα και αναπτυξιακές, ε, αναπτυξιακούς φορείς αλλά και επιχειρήσεις. Υπάρχουν επίσης πολλοί άλλοι δημόσιοι φορείς όπως είναι η Αυστριακή Αναπτυξιακή Τράπεζα που επίσης ε, στηρίζει την επιτέξη των στόχων ε, του θεματολογίου του 2031. 1,2 δις δώσαμε το 2015 ως αναπτυξιακή βοήθεια. Βέβαια, δεν είμαστε στο 0,7% αλλά είμαστε έτοιμοι να βελτιώσουμε την συμμετοχή αυξάνοντας το ποσοστό Επίσης, ε, από τα 5 φτάσαμε στα 20 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Τετραπλασιάσαμε δηλαδή το ποσό. Και σε άλλες περιπτώσεις επίσης έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό. Το 2017 84 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει και δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στον υπαριθμό 6 στόχο που είναι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και θα έχουμε και την Προεδρία ε, της Ένωσης, ε, θα αναλάβουμε πολλά μέτρα σχετικά. Είδαμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί τελευταία στην ε, Ουγκάντα. Και εμείς αναλάβαμε ως περιβα... αναπτυξιακός οργανισμός της αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσουμε τις σχετικές προσπάθειες. Ευχαριστώ. Thank you so much. Now I give the floor to... Ευχαριστώ. το λόγο. Ευρωβουλευτής από το Νόμα των Πρασίνων. Χάιντι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα την παρουσίαση του Ιδρύματος Μπέρτελμαντς. Και ιδίω ένα σημείο με ενδιαφερίδα και τι γίνεται στις σκανδιναβικές χώρες. Οι τέσσερις πρώτες χώρες στο δίκτυ για τους βιώσιμους τόσο ανάπτυξη ήταν από τις σκανδιναβικές από τη Σκανδιναβία. Και ίσως αυτό αποδεικνύει γιατί το σκανδιναβικό μοντέλο είναι ένα ελκυστικό κοινωνικό μοντέλο. Στην επόμενη διαφάνεια όμως είδαμε ότι οι πλούσιες χώρες, που ανήκουν βέβαια αυτές τις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, έχουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις, αυτά spillover. Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Πώς προκύπτει αυτό το αποτέλεσμα. Και το δεύτερο σχόλιο. Η κυρία Πέντους ε, Ρωσιμάνους μίλησε για την εταιρική ευθύνη. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να προσκαλέσουμε τον ιδιωτικό τομέα να συνεισφέρει, θα πρέπει να απαιτήσουμε λογοδοσία από τις επιχειρήσεις. Και εσείς κυρία Πρόεδρε ξέρετε πολύ καλά, ίσως καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι αγώνα δίνουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειάζονται υποχρεωτικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις για την εταιρική ευθύνη, την λογοδοσία σε ό,τι αφορά τα εργασιακά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία εργαζομένων. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών στηρίζει τη γραμμή αυτή. Θα ήταν όμω ενδιαφέρον να ακούσω αν η ίδια συζήτηση γίνεται και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Σε ευχαριστώ Χάιντι και τώρα Αλίου Ακίλα από την Ιγυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Ξένα Ταμάλιο Μολακή λέγομαι, είμαι από την Ιγυρία. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι μπορεί να μην το γνωρίζετε όλοι. Η Ιγυρία έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό, έχει πολύ μεγάλο δυναμικό αλλά και πολύ μεγάλες προκλήσεις ε, στην περιοχή της να αντιμετωπίσει. Λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, ε, της απερίμωσης, ε, αποψήλωσης των δασών, κρίσης εθνικής ταυτότητας, έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Αν δείτε όμως το πρόγραμμα το αναπτυξιακό, UNDP δηλαδή, θα δείτε επίσης ότι πραγματικά πληγωτόμαστε και από πάρα πολύ ψηλά επίπεδα φτώχειας. Πριν από δυόμιση χρόνια αποκτήσαμε ένα νέο ηγέτη που εξηγήνε τα πράγματα στην ε, Νιγηρία σε ό,τι αφορά την καιρό του χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Και γι' αυτό έχουμε και καλή διακυβέρνηση. Η φτώχεια και τα σχετικά εγκλήματα. Μόνο με τη χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να τα αντιμετωπίσει και με μη ισχυρή ηγεσία. Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, έκανε τεράστιες αλλαγές στο μέτωπο της διαφθοράς. Επειδή έγινε λόγος και για φυγή κεφαλαίων και υπόθηκε ότι αυτό πλήττει τα αναπτυσσόμενα κράτη. Αυτό προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε, να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά με σχετική νομοθεσία και με την ε, απονομή δικαιοσύνη. Επίση οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε ένα σχέδιο ανάκαμψης από το 2017 στο 2020 και στόχος είναι η αναγέννηση της ενηγενή οικονομίας. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη, την οικονομική ανάκαμψη, να προωθήσουμε τα παιδιά και, τα, και τις γυναίκες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τονώσουμε την παιδεία, ιδίως ε, την βασική εκπαίδευση. Έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα για την ε, μόρφωση των κοριτσιών, ιδίως από το βορρά. Έχουμε πολλά κορίτσια που δεν πηγαίνουν σχολείο. Επίσης, δίνουμε κάποια μηνιαία υποτροφία και έχουμε και άλλο πρόγραμμα που λέγεται JEEP και έχει στόχο κυρίως τις γυναίκες πάλι. Στόχος μας είναι η κρίση της στόχης όπως σας είπα. Και μας Ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2016 αλλά και το 2017 και 2018 προβλέπει 100 δις ε, του τοπικού νομίσματος ε, για την στέγαση και θα έχουμε μια σύμπραξη μεταξύ κυβέρνηση και ιδιωτικών ε, επιχειρήσεων για να παρασχεθούν ε, προσιτές ε, οικονομικά κατοικίες στους φτωχούς συμπολίτε μας. Ως κοινοβούλιο εργαζόμαστε κι εμείς και το λέει και το Σύνταγμα ότι πρέπει να φτιάξουμε νόμους για τη χρηστή διακυβέρνηση, για την κοινωνική και οικονομική ευημερία των Ιγυριανών. Και εμείς ελέγχουμε τους λογαριασμούς όλων των ε, φορέων και της εκθέσης οικονομικής κατάστασης. Έχουμε επιτροπής, έχουμε την Εθνοσυνέλευση, έχουμε και τη Γερουσία, δύο σώματα. Παρακαλώ μπορείτε να ολοκληρώσετε λέει πρόεδρος. Μάλιστα. Στόχος του Κοινοβουλίου και των δύο σωμάτων είναι να ελέγχουμε τον προπολογισμό την, ε, να εφαρμόζουμε την νομοθεσία και βέβαια πάντοτε σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διαφόρους χορηγούς προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους μας για να βοηθήσουν και αυτοί όσο μπορούν στην εκρίζωση της στόχιας. Thank you. And I give the floor to Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μόνικα Μπάρτος από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που ε, μου δίνετε να μιλήσω. Είμαι Ουγγαρέζα Ευρωβουλευτής. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση για να μπορέσουμε σε αυτό εδώ το κύκλο να σας μεταφέρουμε και τη δική μας εμπειρία. Είμαι μέλος Επιτρόπης Εξωτερικών Υποθέσεων και της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Συχνά λοιπόν παρευρίσκομαι σε τέτοιες ε, εκδηλώσεις και πραγματικά θεωρώ ότι τα εθνικά κοινοβουλιά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν. Είμαστε εκπρόσωποι των ε, πολιτών εμείς οι βουλευτές. Είμαστε οι ενδιάμεσοι, οι διαμεσολαβητές μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Και εμείς πρέπει να μεταφέρουμε τις βασικές ιδέες ε, και τους βασικούς ε, στόχους και προσδοκίες των πολιτών. Και τους στόχους μας μπορούμε να τους πετύχουμε αν εργαστούμε από κοινού με την κοινωνία, από κοινού με τους συνανθρώπους μας. Υπάρχει επίσης ε, πολλής λόγος για την κρίση και για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την επιβάρυνσή του. Πράγματι, Υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν στόχοι. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε να υπάρξει μετάβαση προς ε, μια βιώσιμη ανάπταξη. Και αυτό για να το πετύχουμε πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η απεισόδοξη δεν βοηθάει σε τίποτα. Πρέπει με χαρά να ταινίζουμε το μέλλον, ε, να ενθαρρύνουμε, να εμψυχώνουμε. Και είναι πολύ καλό να ανταλλάσσουμε εμπειρίες, γιατί όλοι έχουμε τις εμπειρίες μας σε ό,τι αφορά και φυσικές καταστροφές και κρίσεις. Θα ήταν πολύ καλό και ευτυχές να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, για ε, τα διάφορα κράτη-μέλη. Είχαμε ε, οργανώσει θα οργανώσουμε μάλλον ένα συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχουν χώρες από την Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και την Αδριατική. Εμείς ε, ως Ούγγροι θα συνεισφέρουμε ε, με μία αναφορά για τα θέματα του ύδατος ε, τη υδάτινης οικονομίας, καθαρισμό υδάτων, επεξεργασία υδάτων. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουμε μπει και νομίζω ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε Όλοι πρέπει να δούμε στις πατρίδες μας τι μπορούμε να συνεισφέρουμε, ποιο λιθαράκι μπορούμε και εμείς να βάλουμε, τι μπορούμε να προσφέρουμε για να βοηθήσουμε ε, και ως Εθνικά Κοινοβουλία. Ευχαριστώ πολύ που δώσετε το λόγο. Now I give the floor to... Ε, Δώστε λόγο στον κύριο Ενρίκη Γερέρο, που είναι και μέλος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, γιατί δεν θα ήθελα να στερήσω χρόνο από τους εθνικούς βουλευτές, αλλά ε, σήμερα συνειδητοποιώ ότι συζητάμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τους επιτύχουμε σε κάθε μία από τις χώρες μας και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε μια εθνική στρατηγική η οποία θα θεμελιώνει την εσωτερική αλληλεγγύη για την επίτευξη του κοινού στόχου. Ε, δεν ήθελα όμως να χάσω την ευκαιρία ως ε, μόνιμος συζητητής για την ανθρωπιστική βοήθεια του Κοινοβουλίου να διαβιβάσω στους εθνικούς ε, βουλευτές τη δραματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο ζητώντας την αλληλεγγύη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 52 εκατομμύρια άνθρωποι ε, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη στιγμή. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πρόσφυγες, εκτοπισμένοι εσωτερικά στη χώρα τους, άνθρωποι που κάνουν αίτηση ασύλου, εκτοπισμένοι επίσης ε, και στην ίδια τους την Ήπειρο και θεωρώ ότι είναι θετικό το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να προβληματιστούμε ε, για κάτι που για μας ήταν ε, ε, πραγματικά μια κρίση που δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Είχαμε απλώς ένα εκατομμύριο ανθρώπους, ενώ για παράδειγμα στο κέρας της Αφρικής αυτή τη στιγμή 20 εκατομμύρια άνθρωποι ε, βιώνουν κρίση και υπάρχει κρίση πείνας και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η επίτευξη των στόχων ε, της ανάπτυξης είναι εσωτερική ανάγκη αλληλεγγύης, αλλά πρέπει να επιδείξουμε και αλληλεγγύη ε, για αυτούς που στον κόσμο ζουν σε μια δραματική κατάσταση, πολύ χειρότερη από εμά και αυτή είναι μια δέσμευση την οποία θα πρέπει να αναλάβουν και τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι Εθνικές Κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πισεγό από την Γαλλία. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ντανιέλ Πισχό, μέλος του Γαλλικού Κοινοβουλίου, μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πελοδομίας. Θα έχουμε υποστηρίξει του θεματολόγιο για το 2030, την καταπολέμηση της φτώχειας, την καταπολέμηση της ε, ανισότητας και όπως πολύ σωστά είπατε όλοι πρέπει να συμμετέχουμε όλοι οι πολιτικοί ε, παράγοντες στη Γαλλία συμμετέχουν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήδη από τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι η εταιρική μας σχέση έχει τεράστια σημασία για την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο, γιατί δεν είμαστε ένα απομονωμένο νησί στον κόσμο, αλλά έχουμε σχέσεις με τους γειτονές μας. υπάρχει από, τις, από την αρχή του το 2010 ε, μια μείωση των διαθέσιμων πόρων για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία, αλλά ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί ότι θα αντιστραφεί αυτή η τάση και θα φτάσουμε στο 0,7% όπως έχουμε δεσμευτεί μέχρι την επόμενη χρονιά. Θα προσπαθήσουμε το Φεβρουάριο ε, του 2018 να ε, αξιοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε μια ε, διυπουργική επιτροπή που θα εξετάσει τα θέματα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Θα προσπαθήσουμε να συμμετάσχουν στη διαβούλευση όλοι οι εμπλεκόμενοι και η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως πάντα. Από την πλευρά μας, ως Γαλλικό Κοινοβούλιο, το Σεπτέμβριο του 2017, οργανίσαμε μια στρογγυλή τράπεζα συζήτησης για το θέμα αυτό στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Το ίδιο πράττει και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα αρμοδιότητάς της. Και όλοι, όλες αυτές οι επιτροπές προσπαθούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε όλη ευθύνη να συνεργαστούμε γιατί μόνο έτσι θα επιτύχουμε τους στόχους που θέσαμε. Σας ευχαριστούμε. Θα δώσω το λόγο στην Λίνα. Όχι, δεν θέλει το λόγο η κυρία Μακάβαν. Θα περάσω στον επόμενο μιλητή. Μαρία Άντερσον από τη Σουήδια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνώ με την συναδελφό από την Νορβηγία το πόσο απαραίτητο είναι να έχουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση της φτώχεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκοσμίω. Χρειάζεται για να συμβεί αυτό να υπάρχουν ε, δίκαιε συνθήκες εργασίας και δίκαιο εμπόριο. Η κοινή αντίληψη, η ευρωπαϊκή για την ανάπτυξη, είναι ένα θετικό βήμα Προ την ανάληψη των ευθυνών που μα αναλογούν για να πετύχουμε το θεματολόγιο 2030. Όμω τώρα πρέπει να δούμε που βρισκόμαστε και τα εθνικά κοινοβούλια να ασκήσουν πίεση στι κυβερνήσει του, καθένα, έτσι ώστε να ε, αναλάβουν τις ευθύνες τους να πράξουν αυτό που υποσχέθηκαν. Ξέρουμε που δεν τα καταφέραμε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Ε, δεν τα καταφέραμε εκεί όπου υπήρχε πόλεμος και δεν τα καταφέραμε όσον αφορά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. υπάρχουν πολυμερείς οργανισμοί, διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΙΕ, όπως η Παγκοσμία Τράπεζα ε, και στο πλαίσιο αυτών συζητούνται τα προβλήματα αυτά. Προσπαθούμε να συζητούμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου του Σουηδικού ε, τα προβλήματα αυτά με σουηδικές με κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα. Έχουμε επίσης ε, στη Σουηδία μια στρατηγική την οποία καταρτίζει η κυβέρνηση και την οποία εφαρμόζει η ΣΥΝΤΑ, η Υπηρεσία για την Αναπτυξιακή Συνεργασία στη Σουηδία. Και αυτέ οι στρατηγικέ έχουν επαναπροσανατολιστεί με βάση του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τι ιδιαίτερα μη αναπτυγμένε χώρε, αναπτυσσόμενε χώρε, και πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα δικαιώματα και στην προστασία των ατόμων με αναπηρία. Θα αναφέρω κάτι που είπε ένα συνάδελφος στην προηγούμενο πάλι, ε, στο προηγούμενο πάνελ, συγγνώμη, ότι ο στόχος που μας αναλογεί εμάς, η ευθύνη που μας αναλογεί εμάς είναι να υποστηρίξουμε ε, τους στόχους κυρία Τελανσουάνα από την Ιταλία, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σταθώ και πάλι στη συζήτηση για τη μετανάστευση. Γιατί η μετανάστευση Πολύ ωραία θα ήταν να μπορούν να εργάζονται όλοι εκεί που ζουν, αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν και ξέρουμε ότι δεν είναι κυβέρνηση στη δυνατή ε, λύση, ε, διότι υπάρχουν και μεγάλες ανισορροπίες μεταξύ ε, φτωχών και πλούσιων χωρών. Στην πραγματικότητα η μετανάστευση είναι ένα από τα πιο μεγάλα στοιχεία ανάπτυξης. Η συμβολή των μεταναστών ήταν πέρσι 500 δις δολάρια, δηλαδή το διπλάσιο των πόρων που δίνουν οι πλούσιες χώρες στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Και πρόκειται για χρήματα τα οποία δεν περνούν από τα σκοτεινά φίλτρα της διαφθοράς, διότι πηγαίνουν απευθείας στις οικογένειες. Και ουσιαστικά η μετανάστευση μπορεί να μετριάσει και την, μετανα... την ανεργία και την υποαπασχόληση στις φτωχές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε το σθένος να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και με μια ρεαλιστική ε, και πιο επιστημονική προσέγγιση και να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για μετανάστευση αναφερόμαστε και σε ανάπτυξη. Δεν αναφερόμαστε μόνο σε επίγωσα κατάσταση και σε απερίμωση χωρών πολλές ευρωπαϊκές χώρες και πολλές περιοχές των ευρωπαϊκών χωρών ε, βγαίνοντας από την κρίση έχουν μεγάλη έλλειψη εργαζομένων και ταυτόχρονα και δραματικές ε, διαδικασίες γύρανσης του πληθυσμού. Η Ιταλία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί στο θέμα αυτό τα τελευταία τρία χρόνια έκανε πάνω από 400.000 διασώσεις στη θάλασσα και προσπαθεί να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα την κρίση στη Λιβύη που πρέπει να πω και την πραγματικότητα ότι την έχουν εγκαταλείψει και οι υπόλοιπε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που ζητώ λοιπόν από όλου είναι να έχουν το σθένος να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα, να μην ε, θεωρήσουν ότι είναι θέμα ταμπού ε, διότι μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ψήφων ε, είναι ένα θέμα το οποίο εάν δεν το αντιμετωπίσουμε θα βρεθεί ε, μπροστά μας στη συνέχεια. Πρέπει λοιπόν ε, να... Ε, ε, δουλέψουμε σωστά, διότι μια πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υλοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν συνεπείς ε, μεταναστευτικές πολιτικές, οι οποίες ε, δεν θα βρίσκουν κάθε χώρα μόνη τους και θα προσπαθεί να δουλέψει μόνη της. Νομίζω η Ιταλία προσπαθεί να κάνει αυτό που της αναλογεί στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το λόγο στην Άννα Τερών από την Ισπανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ισπανία υπάρχει νόμος συνεργασίας και στο άρθρο 15 αναφέρεται στη σημασία των κοινοβουλίων κυρίως στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών. Και λαμβάνοντας υπόψη ε, τη δική μας την νομοθεσία, ε, εντός της ε, Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίες έγινε μια συνάντηση με την κοινωνία των πολιτών και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται απευθείας όχι μόνο με το θέμα της συνεργασίας, αλλά και με τους ε, στόχους της ε, ανάπτυξης που δεν είναι, ε, υπενθυμίζω, μόνο θέμα συνεργασίας. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι θα χάσουμε χρόνο και πρέπει να υπάρχει χρόνος και για τους υπολείπους. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση για το πόσο σημαντικό είναι να λογοδοτεί κάποιο ενώπιον του Κοινοβουλίου, όχι μόνο ενώπιον της Επιτροπής, αλλά ενώπιον του Κοινοβουλίου, διότι το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι το όργανο παρακολούθησης και ελέγχου τη υλοποίησης των πολιτικών της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό το επισημαίνουμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ε, συντάσσουμε ένα κοινό ψήφισμα το οποίο θα υποβάλουμε στο Κογκρέσο των Βουλευτών και η προτεραιότητα στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ε, είναι η πολιτική ε, της κυβέρνησης, ε, διότι οι στόχοι του 2030 είναι οριζόντιοι, δεν θα μπορούν να εξαντληθούν μόνο ε, στην ε, συνεργασία για την ανάπτυξη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όλο το Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε αυτές τις εργασίες, κυρίως οι επιτροπές που είναι κλειδί, επιτροπές για την υγεία, για την εκπαίδευση, για το περιβάλλον, ακόμα και για την οικονομία που είναι θεμελιώδη. και αυτή. Και επίσης ε, νομοθετικές αλλαγές, όπως για παράδειγμα η νομοθεσία για τη συνεργασία τη Ισπανία και οι νόμοι για τι εξωτερικέ σχέσει τη χώρα και νομίζω το έλεγε και ένας ε, συνάδελφος εδώ, τα κοινοβούλια πρέπει να είναι ζωντανά, συμμετοχικά, ανοιχτά και όχι μόνο για το υπόλοιπο κοινοβούλιο, για τις υπόλοιπες χώρες, αλλά και ανοιχτά προς την κοινωνία των πολιτών που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά, διότι εργάζεται απευθείας με τα θέματα αυτά επί και κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να επενθυμίσω. Αυτός ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι μόνο για το δημόσιο τομέα, είναι στόχοι και για τον ιδιωτικό τομέα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στις πολιτικές μας. Δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Και απλώς να υπενθυμίσω ότι δεν μπορούν να είναι απλώς μια μεμονωμένη κίνηση. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά ώστε να μπορέσουν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τα κινεβέλια και να συμμετέχουν ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα, μία απλή ωραία συνάντηση. Πρέπει να ε, οδηγήσουμε σε αποτελέσματα. Έχουμε το καθήκον να υλοποιηθούν όλα αυτά και να είναι πραγματικά. Διότι ε, επήγει σε κοινωνικό επίπεδο το θέμα, γιατί αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Τερών και να δώσω το λόγο στη Μαριέτα Τιρέη από την Ιταλία τελευταία. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής ε, για αυτή την τόσο σημαντική ευκαιρία ε, συζήτησης με διαφόρους βουλευτές. Εγώ, σε συνέχεια των όσων ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες, θα ήθελα να αφαιρθώ στη συμβολή του Ιταλικού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η Ιταλική Γερουσία το Μάιο του 2016 ενέκρινε ψήφισμα για την ανάπτυξη και η καινοτομία είναι το θέμα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Είναι σύνθετο θέμα που χρειάζεται όμως ε, πολιτικές απαντήσεις που δεν θα είναι απλώς κατεπίγουσας ανάγκης. Υπάρχει ε, συμφωνία σχέση σε θέματα μετανάστευσης και το καταπίστευμα για την Αφρική και θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός ε, με δράσεις για την ενόπια των χωρών εταίρων και χωρών καταγωγής και χωρών διέλευσης και θα πρέπει να έχουν και κατάλληλους πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ε, μιας αντιμετώπισης η οποία θα έχει στο προσκήνιο μόνο την ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε κατάλληλα μεθοδολογικά πρότυπα και να δούμε τα θέματα της οικονομίας και της μετανάστευσης. Κατά την άποψή μας, ε, πολλές φορές ανεχτήκαμε την παρουσίαση ε, ε, των πεταναρλιστικών σχέσεων, το Pacta Sunt Servanda, το γεγονός δηλαδή ότι επιτρέψαμε σε κάποιες χώρες να, μην, να αναλάβουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για τους πρόσφυγες. Θεωρούμε ότι είναι επιτυχία του Κοινοβουλίου το γεγονός ότι δόθηκε ελεύθερο φως ε, πράσινο φως για την αναθεώρηση της ε, Συμφωνίας του Δουβλίνου για να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα μετεγκατάστασης όλων των ε, προσφύγων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά επομένουν ακόμα πολλά. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο υλοποίησε ένα πολύ σημαντικό στόχο, τον οποίο προσπαθούσε να υλοποιήσει εδώ και 20 χρόνια, τη μεταρρύθμιση τη εθνική νομοθεσία στη συνεργασία για την ανάστευση, από την οποία δημιουργήθηκε η σύσταση μια Επιτροπής για την ε, Βοήθεια για την Ανάπτυξη και υπάρχουν πολιτικές στις οποίες ασκεί το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων. Το Ιταλικό σύστημα έχει δυναμικές ε, πολιτικές αυτή τη στιγμή, σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικό τομέα και μια πολιτική που θέλει να μειώσει την κατασπατάληση πόρων και να έχει μηχανισμού, συντονισμού αναθέμα και αναγεωγραφική περιφέρεια. Και η Ιταλική κυβέρνηση ανέστρεψε λοιπόν τις τάσεις για τη διαχείριση των φόρων για την βοήθεια για την ανάπτυξη και δίνει όλα ένα και περισσότερους πόρους και βελτίωσε την απόδοση της Ιταλίας για το στόχο του 0,7% του ΑΕΠ. Πόρο απέχουμε βεβαίως ακόμα, αλλά έχουμε αυξήσει και σε απόλυτες τιμές και σε ποσοστά τα ποσοστά. Περάσαμε από τα 2 δις το 2015, είμαστε στα 4,5 δις ε, το 2016 και για ένα σημείο για την Αφρική, η ανάπτυξη της Αφρικής είναι στρατηγική σημασία για την Ιταλία γιατί είναι γέφυρα και σε γεωγραφικό επίπεδο με την Ιταλία και πρέπει να αποφύγουμε την ε, ε, ανασφάλεια και τη δημιουργία της μετανάστευσης. Η Ιτάλα συνέφερε ε, συνεισέφερε στο καταπίστευμα και στη διάσκεψη της Βαλέτας και προώθησε μια νέα συμφωνία με την Αφρική για τη διαχείριση και τη μείωση των μεταναστευτικών ροών, το μεταναστευτικό σύμφωνο. Το 2017 με την νομοθεσία συστήθηκε ένα καταπίστευμα για την Αφρική για 200 εκατομμύρια ευρώ και αυτές τις μέρες εξετάζεται στο Κοινοβούλιο ο προπολογισμό του 2018 όπου θέλουμε το Ταμείο για την Αφρική να γίνει διαρθρωτικό ταμείο με στρατηγικό στόχο η Ιταλία να συμβάλλει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου και να μπορέσει και με αυτό ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε οι Ευρωπαίοι εταίροι να συμμετέχουν και να αυξήσουν και αυτή τη συνεισφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ σύντροφοι και συντρόφισσες για τις παρεμβάσεις σας, για τη συνεισφορά σας σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Για να ολοκληρώσω εγώ προσωπικά και πριν δώσω στον συναρφό μου το λόγο, θα ήθελα απλά και μόνο να πω ότι σίγουρα είναι οικουμενική αυτή η στόχη που αναψάρα και στις αναπτυγμένες και στις αναψώμενες ε, χώρες έχουν υποχρέωση, όπως και ο ιδιωτικό αλλά και ο Δημόσιο τομέα, έχουν υποχρέωση. Έχει ανοίξει ένας δρόμος. Πολλές φορές αυτή η άναρχη παγκοσμιοποίηση και οι ελεύθερες συναλλαγέ μπορεί να οδηγούν το... Ε, σε φαινόμενα τιμωρησίας, ιδίως στι μεγάλες πολυεθνικέ. Ιδίως ε, απέναντι σε συμπεριφορέ και δράσεις ε, που καταπατούν τα εργασιακά δικαιώματα. Έχουμε και για τα... την εξόριξη μεταλλευμάτων και πολύτιμων λίθων από χώρε ε, που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση. Έχουμε θέματα, έχουμε για το φινικέλαιο, για την Global Value Chain, για την εταιρική ευθύνη. Πολλές εκθέσεις έχουμε που βοηθούν για τη βελτίωση της κατάστασης ε, και πολλές εθνικές ε, πρωτοβουλίες όπως από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση που στις αρχές του έτους ένα πολύ σημαντικό νόμο για την εταιρική ευθύνη. Έχουμε και το New Labour Act στη Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία, Γερμανία έχουν σχετικές, ε, σχετικά νομοθετήματα προωθήσει. Άρα άνοιξε ένας δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε και σε συνεργασία ε, μεταξύ μας για να έχουμε αποτελεσματικά επίπεδα ανάπτυξης. Για να κλείσει το δεύτερο με αυτή τη συνάντηση θα ήθελα να σας παρουσιάσω το φίλο και συνάδελφο Άρνε Λίτς, μέλος ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι αρμόδιος για τη σχέση με το Εθνικό Κοινοβούλιο και θα κάνει κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Dear colleagues, it has been... Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν πολύ μεγάλη χαρά μας που σας είχαμε μαζί μας σήμερα στην πολύ σημαντική αυτή συνεδρία για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και για την κοινή αντίληψη, τη συνένεση και χαιρόμαστε πολύ που δεν μίλησαν μόνο ευρωβουλευτές αλλά και συνάδελφοι από την Αφρική που μίλησαν και μας έδωσαν τη δική τους ε, εικόνα της κατάστασης. Να μπορούσαμε να είχαμε λάβει συμμετοχές και από άλλες επίρους ε, και να είχαμε διευρύνει το πλαίσιο. Θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε η συνάδελφο από την Ουγγαρία. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σημαντικό αυτό μονοπάτι που έχουμε ανοίξει μαζί. Πολλοί συνεργάζονται μεταξύ τους και επειδή το είπαμε και στο πλαίσιο της συνένεσης, τα οικονομικά ζητήματα είναι ακρογωνίως λήθος και το, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχει πραγματικά με νόμο κατοχυρώσει το 0,7% είναι κάτι πολύ θετικό. Να δείξουμε ότι το Κοινοβούλιο πιέζει για 0,7%. Και έτσι θα διατηρηθεί και η ισοδοξία τη Ουγγαρίζα ε, συναδέλφου. Ελπίζουμε να φτάσει και η Ουγγαρία στο 0,7%. Με πρόταση πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερε προσπάθειε. Νομίζω ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε ή τέλο πάντων επανασχεδιάσουμε την αρχιτεκτονική τη επίσημη ανεπτυξία βοήθεια. Γιατί το 07 περιλαμβάνει και τη χρηματοδότηση για του μετανάστε. Δεν είναι σωστό αυτό όμω. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Και θα πρέπει το Κοινοβούλιο και τα Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά να ε, κάνουν ό,τι μπορούν η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί ε, στη Γερμανία ε, και ίσως θα πρέπει να πω ένα συγγνώμη εκ μέρους της Γερμανίας γι' αυτό. Πάντως έχουμε μια επιτροπή στη Γερμανία, περιλαμβάνει και ε, μη κυβερνικέ οργανώσεις. Δεν είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό υπάρχει σε άλλες χώρες όπως η Ρουμανία. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο ακόμη πρέπει να μάθει ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να το αντιμετωπίζει μια μεμονωμένη επιτροπή, αλλά πρέπει να σπάσουν κάποια στεγανά και να γίνει μια διακοινοβουλευτική ε, προσέγγιση να υπάρξει. Επίσης μαθαίνουμε και πώς και άλλες επιτροπές μπορούν να συνεισφέρουν. Θέλουμε επίσης μια αντίδραση και από την Κομισιόν με τον κύριο Μίμητσα, Τίμερμανς, ε, την κυρία Μογκερίνη στη Νέα Υόρκη. Ε, είδαμε και είπαμε, δεν υπάρχει ακόμη μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία ουσιαστικά ε, έχει κάνει τη στοχοθέτηση. Θα πρέπει όμως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει περισσότερο. Άρα και εμείς μαθαίνουμε ακόμη εδώ. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει. Το 2019 στη Νέα Υόρκη θα υποβάλουμε την αναφορά μας. Όλοι. Άρα μέχρι τότε πρέπει να καταβάλουμε σκληρές προσπάθειες για να είμαστε επιτυχείς. Από το Ίδρυμα Μπέτερνας είδαμε κάτι πολύ ενδιαφέροντες πίνακες ε, και θέλω να ευχαριστήσω τον Κουίντο. Επίσης ε, η Εστονία μαζί με τη Δανία παρουσίασε Πώ ε, οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη και κλωση πηγαινουν πηγαίνουν χέρι-χέρι. Θέλω να ευχαριστήσω την Εστονική Προεδρία. Η Λόλα επίση έχει κάνει μια έκθεση για μια πρωτοβουλία για τον τομέα τη ένδυση των υφασμάτων, τη κλωστοϊφαντουργία. Και είναι εμβληματική πρωτοβουλία. Έχουμε ήδη πρόοδο σε Δανία, Γερμανία, Ολλανδία. Υπάρχει μια στρατηγική στι χώρε αυτέ για μια πιο βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού σε υφάσματα. Ζητούμε οι Επίτροπή μας να αναλάβουν πρωτοβουλίες και καλό θα ήταν επίσης και σε επίπεδο ΙΕ μέσω των στόχων βιώσιμης αλλά και όλοι οι συνάδελφοι να βοηθήσουμε για την κλωστοϊφαντουργία, φαντουργία για τα υφάσματα. Και αν μπορούμε θα σας δώσουμε ε, τις σχετικές πληροφορίες ε, για να προωθήσετε το θέμα στα εθνικά σας κοινοβούλια. Πολλές φορές επίσης έγινε λόγος για τη σημασία του κλίματος, το είπαν οι συνάδελφοι από την Αφρική και για τα εφάσματα. Έχουμε το θέμα της ε, βιώσιμης παραγωγής. Έχουμε και το στόχο 13 για την κλιματική αλλά και άλλες δράσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι μέλλον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Θέλουμε τώρα μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να καταθέσουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για την κλιματική διπλωματία. Προσπαθούμε δηλαδή να συνενώσουμε διάφορα πράγματα από την αιγίδα τη Επιτροπή Ανάπτυξης αλλά και με συνεργασία με άλλε επιτροπέ. Εν ώψη δε της επόμενης ε, συνόδου που θα έχουμε, ήδη σκέφτομαι από τώρα, θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε κάποιε βέλτιστες πρακτικέ. Ήδη ενημερωθήκαμε για κάποιε βέλτιστες πρακτικέ. Θα μπορούσε να είναι ένα από τα σημεία στη μεσιά διάταξη η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από τι δικές σα χώρε για του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη. Τι κάνετε εσεί στο πέστο του κοινοβουλευτικού σα έργου. Υπάρχει διακοινοβουλευτική συνεργασία μεταξύ περισσότερων επιτροπών των κοινοβουλίων σα. Θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε στην ημερήσια διάταξη την επόμενη φορά. Θα ήθελα επίση να σα ανακοινώσω ότι μετά τη συνεδρία αυτή θα μπορέσουμε να τα πούμε. Έχουμε σάντουιτς τα οποία σερβίρονται στην καφετέρια στον τρίτο όροφο, ένα επίπεδο πιο κάτω δηλαδή, έναν όροφο πιο κάτω, εδώ στο κτίριο που είμαστε και εκεί θα έχουμε μια εξαιρετική ευκαιρία να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις πιο χαλαρά, να μιλήσουμε και με τους προσώπους του Ιδρύματος Μπέρτελ μας, που είναι εδώ και έχει κάνει εκθέσεις για τις χώρες σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και στο βίντεο που έφταξαν το βίντεο που είδαμε πριν. ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας, ε, τους συνεργάτες των Ευρωβουλευτών. Θέλω να σας πω επίσης ότι η Επιτροπή μας συνεδριάζει ξανά στις 3. Το λέω αυτό για τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου. Επίσης, στην αρχή σας ε, είπαμε ότι έχουμε αυτούς τους στόχους έξω, έξω από την αίθουσα, στο δεξί χέρι. Αν θέλετε να φωτογραφηθείτε μπροστά στον πιο σημαντικό στόχο, μπορείτε να πάρετε φωτογραφία, να βάλετε από κάτω ένα quote και να το ανεβάσετε στο διαδίκτυο ή να το στείλετε με ένα email, να περάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα σας στείλουμε και τις πληροφορίες από τον Μπέρτελσμα, θα σας στείλουμε το link για το βίντεο. Θα μπορούσατε να δείξετε στο, Εθνικό Κοινοβούλιο τη χώρα σα και για τη συνένεση στην κοινή αντίληψη μπορούμε να σα στείλουμε πληροφορίε εφόσον το επιθυμείτε. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τι παρεμβάσει σα και θα τα πούμε στον πιο κάτω όροφο στην καφετέρια ή μπροστά εδώ στι φωτογραφίε. Ο πρόεδρο ευχαριστεί και του διερμηνεί που παρέμουν. Thank you. Thank you.